I open our afternoon meeting for today. Ξεκινάμε την απογευματινή μας συνεδρίαση για σήμερα, εφόσον το επιτρέπετε. Δεν είμαστε και πάρα πολύ τώρα εδώ που τα λέμε. Το κύριο θέμα το οποίο θα μας απασχολεί σήμερα είναι η δημόσια κρόαση για την απλοποίηση και την κοπή του, της ερυθρής κορδέλας, δηλαδή της γραφειοκρατίας, στα ευρωπαϊκά διαφορετικά ταμεία και τις επενδύσεις. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το μέλλον και της πολιτικής συνοχής με την πολύπλοκη επιμερισμένη διαχείρισή της. Αυτό θα είναι ένα κέριο θέμα για το νομοθετικό πακέτο ήταν και σημαντικό, για το πακέτο για την ε, περίοδο 2014-2020. Ο στόχο τη απλοποίηση, είναι να βελτιώσει την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής και να αυξήσει την αποδοτικότητα της καθώ και την προσβασιμότητα στα ευρωπαϊκά ταμεία περιφερειακού χαρακτήρα και συνοχής. Έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια πολλέ πρόνοιες για να υπάρξει εναρμόνιση και απλοποίηση των διαδικασιών η μείωση του διοικητικού άχθους για τους δικαιούχου βρίσκεται στον πυρήνα της απλοποίηση. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό, περιφερειακό και φυσικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων <clears throat> είναι ένα από τα κύρια θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Ρέντζη. Γι' αυτό χαίρομαι που μπορώ να υποδεχθώ τέσσερις εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό το πρόγραμμα της ακρόασης έχει διανεμηθεί χωριστά. Το πρόγραμμα υπάρχει στα χέρια σας. Θα δώσω τον λόγο στον πρώτο στους καλεσμένους μας για 10 λεπτά κάθε φορά και μετά στο αμέλη μας για ερωτήσεις και απαντήσεις καθώς και στον εκπρόσωπο της Κομισιόν αν θέλει να κάνει παρατηρήσεις σε σχέση με τα θέματα αυτά. οι καλεσμένοι μας τώρα. Η Αντζέλικα Ποτς Μόγγελε, η οποία είναι αρμόδια για την απλοποίηση στις, στους Δήμους και τις Περιφέρειες, η κυρία Άννα Μαρία Καντέλα από την Απουλία, ο κύριος Γεώργιος Ρης από την Βάδιν Βιρτενβέργιν και ο καθηγητής Βασίλης Ντογκάρου από την Τιμισουάρα στη Ρουμανία. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την Αγγελική Ποθ γέλεν. Έχετε 10 λεπτά για να κάνετε την ε, παρουσίασή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή σα που κάλεσε το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών για να μοιραστούμε μέσα στην εμπειρία μα. Θα σα υπενθυμίσω ο οργανισμό μα. Είναι ο οργανισμός που εκπροσωπεί όλε τι Εθνικέ ενώσεις περιφερειακών και τοπικών ε, αρχών και τα όσα θα σα πω σήμερα βασίζονται σε πληροφορίες που έχω λάβει από συναδέλφου από ενώσεις μέλη που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση των διαφορετικών ταμείων και των επιχειρηματικών προγραμμάτων ε, ε, στις περιοχές τους και εγώ επιλέγει για να παρουσιάσω την εμπειρία μας μέχρι στιγμής. Έχουμε ετοιμάσει κάποια έγγραφα που θα βρείτε στους φακέλους σας, αλλά αν θέλετε άλλε πληροφορίες μπορούμε να σας τις στείλουμε μετά από την ακρόαση. Μια μικρή αξιολόγηση της κατάστασης από την πλευρά μας είναι ότι μπορούμε να πούμε για τους δικαιούχους ένα βήμα προς την απλούστευση έχει επιτευχθεί με την ενιαία προσέγγιση ε, την ηλεκτρονική τεκμηρίωση και την ε, ορθή διαχείριση. Αλλά οι κανόνες εξακολουθούν να είναι υπερβολικά πολύ για τις διοικητικές αρχές. Όσον αφορά την ένταξη των ταμείων, έχει δημιουργηθεί σύγχυση. Οι κανονισμοί που παρέχουν το πλαίσιο για την εδαφική ανάπτυξη, τα CLLD, τα ITI και όλα αυτά ε, τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτά τα κονδύλια επιτόπου και να επισημάνω τέσσερα βασικά στοιχεία για την εναρμόνιση, για την ευελιξία και την ε, αναλογικότητα και τη διαχείριση βασισμένη σε αποτελέσματα. Όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων, ε, η προσέγγιση πολλών ταμείων ε, θεωρείται καλή, αλλά αυτό που είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, όπως γνωρίζετε υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικοί κανόνες, διαφορετικά ταμεία και επιπλέον κάθε κράτος μέλος αυτό ανατεθεί σε διαφορετικά υπουργεία και διάφορες γενικές διευθύνσεις εμπλέκονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε το, η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα περίπλοκη. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε να κάνουμε τις εξής συστάσεις. Τα μέσα τα οποία προτείνονται στους νέους κανονισμούς όπως τα ενδιάμεσα όργανα, η ITI και η CLLD βοηθούν ε, για την απλούστευση αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί ευρέως. Πρόσφατα προέκυψε μια επικαιροποιημένη ε, μελέτη για τις ITI στα κράτη-μέλη και όπως φαίνεται η εφαρμογή είναι αργή. Ε, θέλουμε να ενθαρρύνουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα ευρύτερα διότι πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθούσε να απλούστευση. Θέλουμε να παρακινήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί προς κοινέ διαδικασίες και ως στο βαθμό του δυνατού και πιστεύουμε ότι το ESIF ήταν ένα καλό βήμα αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιο μακροπρόθεσμα θα θέλαμε να προτείνουμε να υπάρχει μια ενιαία ροή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το τοπικό επίπεδο που να αντιμετωπίζω ε, τις διάφορες ε, ε, ανάγκες που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο να είναι μια ενιαία ουσιαστικά υπηρεσία που να καλύπτει όλες τις ανάγκες των ετούντων με μια ενιαία πηγή χρηματοδότηση απευθείας στις περιφερειακές και τοπικές περιοχές με αντάλλαγμα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχουμε προετοιμάσει και κάποια παραδείγματα, αλλά θα τα παραλείψω εδώ τώρα. Το δεύτερο σημείο αφορά την ευελιξία. Η ευελιξία είναι κάτι που ακόμη δεν έχει επιτευχθεί. Η Κομισιόν έχει ορίσει τα θέματα προτεραιότητας και τα ποσοστά εθνικών προγραμμάτων, αλλά από την εμπειριά μας, ειδικότερα τα μικρότερα κράτη-μέλη, δεν έχουν σχεδόν καμία ευελιξία ε, όσον αφορά τις επιλογές τους. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που έχουμε δώσει, το, σα δώσαμε είναι το παράδειγμα των κατοχωρών. Όσον αφορά την αναλογικότητα και το ζήτημα των ελέγχων και των οικονομικών ελέγχων, δεν θα σα εκπληξεί ότι εδώ έχουμε λάβει πολλά σχόλια από τους συναδέλφου μας, όπου αναφέρεται ότι τα διαρθρωτικά ταμεία εξακολουθούν να έχουν πολυεπίπεδους ελέγχους, πολλούς δηλαδή ελέγχους των ίδιων εγγράφων από διαφορετικές αρχές σε διαφορετικά επίπεδα και συχνά έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό δημιουργεί νομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα για τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές αλλά κυρίως και για τους δικαιούχους. Ένα βασικό κριτήριο για την απλούστευση όσον αφορά τους δικαιούχους συμπεριλαμβανομένων των τοπικών περιφερειακών αρχών είναι η μείωση του αριθμού των απαιτούμενων ελέγχων. Ο σημερινός αριθμός ε, θεωρείται υπερβολικός. Ορισμένες χώρες έχουν εθνικές δηλώσεις ε, που συνεπάγονται περισσότερους εσωτερικού ελέγχους και λιγότερους ευρωπαϊκούς ελέγχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τίνει να αυξάνει τους ελέγχους σε χώρες ε, όπου διαπιστώνεται ψηλό ε, ποσοστό σφάλματος από το ελεγκτικό συνέδριο αυτό μπορεί να δημιουργεί δυσανάλογες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών με αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους. Το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι όλα τα κράτη-μέλη ε, είναι ίδια και ότι τα προβλήματα που εμφανίζονται σε μια χώρα εμφανίζονται και σε μια άλλη. Ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει πραγματικά. Οπότε εμείς έχουμε να προτείνουμε το εξή ε, μια πιο αναλογική προσέγγιση βασισμένη σε αποτελέσματα όσον αφορά τους ελέγχους με λιγότερη εστίαση στις ποινές και μεγαλύτερη εστίαση στη βελτίωση θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση πιο προσαρμοσμένη στο κάθε κράτο μέλο και να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ απάτης και σφάλματος. Πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο σύνολο ε, ε, κανόνων ελέγχου, να γίνεται αξιολόγηση κινδύνου σε συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις πρακτικές που να αναπτυχθεί με τη βοήθεια του ελεγκτικού συνεδρίου να υπάρχει μια πιο ελαφριά διαδικασία, εκχωρώντας περισσότερο έλεγχο στι εθνικές αρχές, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις φυσικά, για παράδειγμα, θα μπορούσε να εισαχθεί ένα σύστημα ε, ενιαίας ενημέρωσης ενημέου ελέγχου, single information, single audit, που να έχει θεθεί από όλα τα μέρη, από την Κομισιόν μέχρι τους δικαιούχους. Οποιασδήποτε αλλαγές στους κανόνες ή ερμηνείες των κανόνων που ε, εμφανίζονται στη μέση του προγράμματο δεν μπορούν να εφαρμόζονται αναδρομικά εάν πρόκειται να ε, ε, βασιστώ να επιβληθεί κάποια ποινή ε, στα κράτη-μέλη ή στις διοικητικές αρχές στους τοπικούς δικαιούχους ε, αν θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνονται είναι σημαντικό οι ελεκτικές αρχές να συναντώνται από πρώιμο στάδιο κατά το σχεδιασμό των συστημάτων ώστε να αποφεύγονται αντιφάσεις αργότερα και το τελευταίο θέμα είναι ότι η συμμόρφωση μπορεί να βελτιωθεί μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας των διαδικασιών ελέγχου έτσι ώστε λοιπόν η Κομισιόν μπορεί να δημοσιεύει τα ευρήματα τη πιο νωρί κατά τη διαδικασία. Το τελευταίο σημείο αφορά τη διαχείριση βάσει αποτελεσμάτων. Λέμε ότι είναι κρίμα που η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη έχουν εγκαταλείψει τη δυνατότητα ανάπτυξη κοινών σχεδίων δράση. Αυτά τα κοινά σχέδια δράση έχουν τη δυνατότητα καταπολέμηση τη γραφειοκρατία ε, και των ελέγχων ε, για όλα τα ταμεία αλλά δεν ε, δεν θέλησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τέτοια JAP, τέτοια κοινά σχέδια δράση. Ουσιαστικά η καθοδήγηση δίδεται συχνά πολύ αργά και δεν είναι σαφής. Όπως γνωρίζουμε στη σημερινή προγραμματική περίοδο, η Γενική Διευθύνση Ρίτζο ε, έγραψε τι καθηγητήρες γραμμές για τα CLD και τα ITI το καλοκαίρι του 2014 ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει τα προγράμματα του στο κράτη-μέλη συνεπώς ήταν πολύ αργά για να χρησιμεύσουν σε οτιδήποτε οι κατευθυντήρες γραμμές οπότε θα θέλαμε η Κομισιόν να προετοιμάζει τα κατευθυντήρια έγγραφα έγκαιρα. Θα επιθυμούσαμε στο μέλλον η Κομισιόν να ε, παρουσιάζει κατευθυντήρες γραμμές μαζί με τις προτάσεις ε, νέας νομοθεσίας. Αυτό θα κάνει τη ζωή όλων ευκολότερη διότι εκεί η Κομισιόν θα έχει δώσει σαφείς ιδέες για το τι αναμένει από τα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες και τους δήμους. Επίσης και τοπικοί δικαιούχοι ζητούν ε, πληροφορίες για την υλοποίηση των ταμείων, για παράδειγμα όσον αφορά την κρατική ενίσχυση κανονικά οι κατευθύνες γραμμές κομιστών έπρεπε να αρκούν χωρίς να δίνονται άλλες από τις τοπικές αρχές. Ε, ωστόσο, οι κατευθύνε γραμμέ ε, απευθύνονται όλε στι διοικητικέ αρχέ, ε, στου διοικητικού οργανισμού και είναι μόνο στα αγγλικά. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη ανάπτυξη των δυνατήτων σε όλα τα κράτη-μέλη και επίση θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι διαχειριστικέ αρχέ περισσότερο το θεματικό στόχο 11 τα ερωτήματα κλειδιά παραμένουν είναι τι είναι η απλούστευση, μπορούμε να συμφωνήσουμε ενό κοινού ορισμού, ποιο είναι ο στόχο τη απλούστευση, ποιοι θα πρέπει να είναι οι βασικοί δικαιούχοι τη απλούστευση και πώ μπορούμε να επιτύχουμε αυτού του στόχου. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα επωφέλε να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στη διαδικασία προβληματισμού, ώστε να υιοθετηθεί μια ενθαρρυντική προσέγγιση, μια ε, θεραλέα προσέγγιση, συγγνώμη, για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, να εκχωρείται ευθύνη από την κεντρική κυβέρνηση με ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο και στόχους βασισμένους αποτελέσματα. Τέλος, το CMR, ο Οργανισμός ε, Ενώσεων Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, ε, δεσμεύεται να ξεκινήσει μια ε, εποφελή διαδικασία προβληματισμού για να βρεθούν τρόποι απλούστευσης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και της υλοποίησής τους. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Αναμαρία Μαρία Καντέλα για συγκέντρωση και σωμάτωση των ε, νέων ταμείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Ανάπτυξης Υπέθρου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα εμβαθύνω στο ζήτημα της εμβάθυνσης ε, των κανόνων χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων έχοντας επιλέξει να εστιαστώ στον θεματικό στόχο 9 πιο συγκεκριμένα που αφορά το προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αυτός είναι και ο θεματικός στόχος και ο τομέας προγραμματισμού όπου κατά την άποψή μου θα απαιτείται περισσότερη απλούστευση. Είναι ο θεματικός στόχος όπου υπάρχει πολύ σημαντική σχέση, πολύ ισχυρή μεταξύ του καταμερισμού των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου συγκεκριμένα για την καταπολέμηση της φτώχειας και την πριώθηση της, ε, ε, των κοινωνικών θεμάτων και υπάρχει και άλλη μια σχέση σημαντική το να ενταχθούν οι διάφοροι πόροι των ταμείων στον στόχο αυτών. Εγώ στην ε, περιοχή της Πούλια διευθυνώ την υπηρεσία ε, κοινωνικού προγραμματισμού και υγειονομικού προγραμματισμού τα τελευταία δύο χρόνια ε, εργαζόμαστε στην ανάπτυξη του προγράμματος 2014-2020 και είμαστε η περιφέρεια που επέλεξε να αξιοποιήσει στο μέγιστο την ευκαιρία που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη ενός ε, πολυταμιακού προγράμματος ε, στην, ε, στις περιοχές του 2000, μέχρι το 2013 όπου ε, αντιμετωπίζαμε ξεχωριστά τα δύο ταμεία με εντελώς ξεχωριστούς κανόνες αλλά και με ένα προγραμματισμό, με δύο προγραμματισμούς που λειτουργούσαν παράλληλα χωρίς να συγκλίνουν για να επιτευχθούν οι στόχοι ανάπτυξης. Οπότε αυτή η ευκαιρία του πολυταμιακού ε, προγράμματος είναι εξαιρετικά σημαντική. Οπότε αποφασίσαμε να την αξιοποιήσουμε. Βάσει αυτής της εμπειρίας που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια, όπου ε, κάναμε τον προγραμματισμό και τώρα αρχίζουμε την υλοποίηση, θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα σημεία ε, όπου θα πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα η εναρμόνιση των ε, κοινοτικών και εθνικών κανόνων, αλλά και μεγαλύτερη σύγκληση μεταξύ των κανόνων χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των κανόνων ε, της χρήσης ε, του άλλου ταμείου, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, όσον αφορά τα ζητήματα που θα ήθελα να εξετάσουμε εδώ ε, στα γρήγορα. Σίγουρα θα αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε ένα, στο, στο, στην απασχόληση, στην κοινωνική καινοτομία και στην κοινωνική ένταξη χαρακτηριστικό που διέπει όλα πλέον τα προγράμματα της ε, κοινότητα και το ζήτημα τη φτώχεια Επίσης ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι εκείνο που αφορά το σύστημα των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση των στόχων του ε, νέων προγραμμάτων. Ε, οι εμπλεκόμενοι είναι πιο πολυάριθμοι, όχι μόνο αριθμητικά, είναι και, και πολυπίκυλοι περισσότερες αρχές, περισσότερες ενέσεις, ενώσεις από ε, τις ε, τοπικές αρχές μέχρι ιδιώτες, ε, κοινωνικές οργανώσεις, εμπλεκόμενοι στην κοινωνική οικονομία. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο εμπλουτίζεται όλο και περισσότερο. Πρόκειται για ένα σύστημα αξιοποίησης σχέσεων και δημοσιοδιωτικού τομέα με πολύ πιο διαφοροποιημένο και πολύ ποικιλό τρόπο από το τρέχον πλαίσιο κανονισμών και με μεγαλύτερη δυνατότητα αξιοποίησή του. Το πλαίσιο κανόνων κοινωνικού ταμείου και ε, ε, περιφερειακής ανάπτυξης είναι πολύ πλούσιο. Ουσιαστικά βασίζεται σε περιφερειακές ε, δομές που συχνά έχουν εμπειρία εργασιακή και συγκεκριμένα συστήματα διαδικασιών και ελέγχων που απορρέει από την ξεχωριστή διαχείριση των ταμείων. Απορρέει επίσης από έναν ισχυρό ε, διαχωρισμό, απομόνωση των δημοσίων ενδιαφερομένων και των ιδιωτών ε, και κάνει και διάκριση επίσης μεταξύ όσων προωθούν τις παρεμβάσεις και, όσων τις, ε, και των δικαιούχων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του θεματικού στοχονιά για την ενεργό κοινωνική ένταξη και που θα παίξει σημαντικό ρόλο για τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα όπως και για το εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ειδικού μας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών. Ρόλο λοιπόν σημαντικό όπως έλεγα θα παίξουν οι τοπικές αρχές, οι Δήμοι όσον αφορά την Ιταλία. Ε, οι Δήμοι οι οποίοι θα συνενώνονται σε ευρύτερε ε, διοικήσεις ε, πέραν των συνόρων των Δήμων ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη εναρμόνιση. Σε αυτή την περίπτωση οι Δήμοι λοιπόν, οι οποίοι θα είναι δικαιούχοι, θα εργαστούν εν μέρη και για την υλοποίηση ορισμένων από τις παρεμβάσεις. Ε, συνεργάζονται για την επιλογή των, επιχείρη, των δράσεων που θα γίνουν και είναι επίσης και δικαιούχοι και εμπλέκονται επίσης και στην επιλογή και την πολυδιαστασιακή ε, ε, αξιολόγηση είναι ένας ρόλος σημαντικός, ε, ρόλος που καταδεικνύει την ελάχιστη δυνατότητα ε, διαχείρισης όλων αυτών των ε, κονδυλίων στο ύψος των περιστάσεων. Από τη δική μας εμπειρία για την περίοδο 2007-2013 διαπιστώνουμε ότι οι προσπάθειες των διαχειριστικών αρχών για να συνδέσουν τους εθνικούς και περιφερειακούς κανόνες με τους κοινωτικούς σε εγχειρίδια και κατευθυντήρες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων στις αρχές ελέγχου απεφέρει σημαντικά αποτελέσματα και όσον αφορά την κατάρτιση, την εκπαίδευση, την προετοιμασία ε, των ε, όσων ε, κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν τις πηγές χρηματοδότησης διότι αντικειμενικά το να υπάρχουν διαφορετικά πλαίσια κανόνων επειδή προέρχονταν από διαφορετικές αρχές και η σύνδεση αυτών για τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων δεν ήταν κάτι απλό, δεν ήταν κάτι που μπορούσαν να πράξουν ενιαίες επιμέρους διοικητικές αρχές. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι στο μεταξύ οι κατήτερες γραμμές ε, χρησιμεύσαν για την υποβολή εκθέσεων ε, για το κοινωνικό ταμείο, για παράδειγμα για όλα τα προγράμματα κοινωνικών υποδομών, όπου εμείς προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε εκτός από τις, διευθύνσεις, εκτός από τις, γραμμές, από τις γραμμές υποβολής εκθέσεων και για τις ε, διαχειριστικές αρχές και για τις ελεκτικές αρχές τα χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε αυτές τις τέτοιες γραμμές και για τις ε, ε, ελεγκτικές αρχές. Αυτό είναι μια πρώτη προσπάθεια που θα πρέπει να συνεχιστεί σε αυτό το προγραμματικό κύκλο ώστε να δώσουμε, να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι μια δομή ε, ανώτερη η αρχή ελέγχου και οι δραστηριότητες ελέγχου. Θα πρέπει λοιπόν όσοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή να γνωρίζουν τι κάνουν και οι αρχές ελέγχου. Όλο αυτό βοηθά στο να προετοιμάζονται φάκελοι προγραμμάτων που να δημιουργούν λιγότερη σύγχυση, που να έχουν μια πιο ομαλή διάρκεια ζωής, ώστε να απλουστεύονται και οι δραστηριότητες των ελεγκτικών αρχών. Ε, φυσικά για τους ελέγχους υπάρχει και ε, το θέμα της ε, προσαρμογής με τον τύπο του έργου, το μέγεθος του έργου, και το είδος και των δικαιούχων που πρέπει να εφαρμόσουν τα έργα. Το να χρησιμοποιούμε τις ίδιες λίστες ελέγχου για προγράμματα διαφορετικών διαστάσεων και διαφορετικών χαρακτηριστικών και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ε, μη συγκρίσιμων σε σχέση με τον νέο κύκλο προγραμματισμού αρκεί να αναφερθώ στο ε, σημαντική όθηση που έχει δοθεί στο νέα προγραμματική περίοδο στον ευρύτατο τομέα, όπου δεν θα επεκταθώ αυτή τη στιγμή, που είναι ο τομέας της κοινωνικής καινοτομία. Στον τομέα αυτό οι δράσεις θα είναι εντελώς νέες ε, σε σχέση με ε, για τις διάφορες περιοχές με διάφορους βαθμούς πολυπλοκότητας. Το να εργαζόμαστε τώρα με τις ίδιες λίστες ελέγχου σε όλα αυτά τα προγράμματα ε, σημαίνει ότι διατρέχουμε τον κίνδυνο να ε, βαρύνουμε υπερβολικά την ε, διαχειριστική δομή ε, και στο τέλος ε, θα φαίνεται σαν στόχος να ήταν μόνο η σωστή διαχείριση ενώ η σωστή διαχείριση πρέπει να είναι η βάση και όχι ο στόχος θα πρέπει να είναι το κοινό χαρακτηριστικό που θα διέπει όλες μας τις ε, δραστηριότητες ενώ στόχοι μας είναι οι αλλαγές που θα φέρουμε στις διάφορες περιοχές και οι καινοτομίε που θα εφαρμόσουμε πειραματικά στους διάφορους δικαιούχους ειδικότερα Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων που θα προωθήσουμε, ειδικότερα για το στόχο ενεργού κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της στόχες, Η ανάγκη αυτή που μας διδάσκει ότι χρειάζεται συνεργασία ιδιωτικού και ε, δημόσιου τομέα για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι ε, εκεί συμβαίνει το ίδιο όπως και στην καινοτομία, των να πειραματιστούμε με νέες ή ασυνήθιστες μορφές συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ασυνήθιστες ε, στο πλαίσιο αυτών των ταμείων, μέσω συνεταιρισμών, μέσω ε, κοινοτήτων και ενώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές και για να προωθήσουμε την ενεργοϊθαγένεια, τον καταμερισμό των πόρων. Το θέμα του welfare sharing δεν είναι πια μόνο θεωρία οι κοινότητε μας καθημερινά ε, ζουν, ε, βιώνουν εμπειρίες πολύ σημαντικές στον τομέα αυτών. Αν θελήσουμε σήμερα να πλαισιώσουμε όλα αυτά με δύο διαφορετικά συστήματα κανόνων ε, του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου ε, ε, υπάρχει περίπτωση να έχουμε την ανεπιθύμητη αντίδραση από τις περιοχές, δηλαδή να μας δείξουν έλλειψη βούλησης και μετά αποθεάριζε κάποια αντίσταση όσον αφορά την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων. Με πιθανό αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, ξέρετε, η εργαλειοθήκη που έχουμε σήμερα στα χέρια μας μάλλον διαχωρίζει παρά συνενώνει. Το παράδοξο είναι ότι έχουμε ένα πολυταμιακό πρόγραμμα, προσπαθούμε, θα προσπαθήσουμε να ε, αναπτύξουμε δράσεις ε, στο μέγιστο δυνατό βαθμό με δυνατότητα ένταξης και δεν έχουμε ακόμα ένα σύστημα ελέγχου που να επιτρέπει έναν ενιαίο πλήρη έλεγχο των διαστάσεων ε, που χαρακτηρίζουν περισσότερο το κοινωνικό τομέα και περισσότερο το ε, περιφερειακή ανάπτυξη. Να προσθέσω κι άλλο ένα ζήτημα. Εμείς εδώ αναφερόμαστε σε δύο γενικές διευθύνσεις ε, όταν αναφερόμαστε σε πολυταμιακή διάσταση. Έχουμε δύο γενικές διευθύνσεις. Εμείς αναπτύσσουμε τοπικά σχέδια δράσης που περιλαμβάνουν τους διάφορους πόρους ε, μαζί και μετά στη συνέχεια όταν ε, έρχεται ο έλεγχος από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξαφνικά λαμβάνουμε ξεχωριστά τον ελεκτικό συνέδριο που δεχόμαστε, ε, μετά ξαφνικά έρχεται η Κομισιόν, οι οικονομικοί ελεγκτές ε, για τα κράτη-μέλη και ε, μερικές φορές αυτό που είναι πολύ διασκεδαστικό είναι ότι γίνεται δειγματοληψία στα ίδια έργα, στα ίδια προγράμματα. Αυτή η δειγματοληψία που γίνεται επί ενός ε, προγράμματος μπορεί να γίνεται από κοινού για όλους. δηλαδή αφού ελεγχθεί, να ελεγχθεί πλήρως από όλες τις διάφορες ελεκτικές αρχές το ίδιο δείγμα έργου παρά να έρχεται ο καθένα ξεχωριστά κάθε τρει-τέσσερι μήνε ε, και να προγραμματίζει μια άλλη επίσκεψη για μια άλλη αρχή. Εδώ μιλάμε τώρα για αρχές, για ιδιώτες που δεν έχουν κάποια γενικότερη δομή για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων. Έχουν μια ξεχωριστή ζωή και χρειαζόμαστε κάποιο εξορθολογισμό σε μεγαλύτερο βαθμό εμείς στην Ιταλία λέμε αποτελεσματικότητα, φιτσενταμέντο όπως λέει ο Μουλίτρε, αλλά δύσκολο να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Πριν λοιπόν αλλάξουμε, ε, συγγνώμη, εισάγουμε στοιχεία απλούστευση στο σύστημα κανόνων, ε, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να σκεφτούμε το ενδεχόμενο κάποιο εξορθολογισμό των διαδικασιών ε, των διαδικασιών με τις οποίες λειτουργούμε όλοι και φυσικά αναφέρομαι εδώ στι δραστηριότητε φυσικά ενίοτε και των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Δεν αναφέρομαι μόνο στι κοινωτικέ αρχέ. Και με αυτό για να κλείσω έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια και προσπάθεια αλλαγής νοοτροπίας ώστε στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 οι χώρες ε, που δίνουν περισσότερη προσοχή σε ολοκληρωμένους ε, στόχους ε, δεν έχουν προγραμματίσει όλες οι χώρες ένα προγραμματισμό με ένα μέσο με ένα μονοταμείο εμείς όμως έχουμε επιλέξει ένα πολυταμιακό πρόγραμμα εμείς ζητάμε οι προσπάθειες εφαρμογής τουλάχιστον κατά το πρώτο διάστημα βάσει του σημερινού, των σημερινών κανόνων που έχουμε αυτό που λέμε ότι υπάρχει κίνδυνος να κινηθούν σε όλα αυτά σε παράλληλες τροχές που δεν θα οδηγήσουν απαραίτητα σε αποτελεσματική διαχείριση παρά τις προσπάθειες που εμείς ε, προσπαθούμε να καταβάλουμε ως διαχειριστικές αρχές ώστε να μειώσουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό που οφειλέται σε αυτούς τους κανόνες που μας επιβάλλονται από τις άλλες αρχές. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κάπως ε, υπάρχει μια πίεση χρόνου βέβαια. Πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο μας. Θα δώσω το λόγο τώρα στον επόμενο ομιλητή μας. George ε, Rich, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του ΙΕΦΡΕ από την Βάδιν και Βιρτεμβέρη, του Περιφερειακού Ταμείου από την Βάδιν Βιρτεμβέρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω και τη δική μας έτσι, άποψη των δημόσιων υπαλλήλων, των διοικητικών αρχών. Να σας δώσουμε λοιπόν και την άποψη της βάσης της διοίκησης. Θεωρώ πως το ταμείο ε, γεωργικής ε, ανάπτυξης και τα περιφερειακά ταμεία δεν μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Αντίθετα μας κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη. Καταρχάς, να σας πω δύο λόγια για τον εαυτό μου. Είμαι από την Στουτγάρδη, είναι αυτό το μικρό κίτρινο σημείο στο χάρτη. Αν δεν ξέρετε που ανήκει η Στουτγάρδη και ποια είναι η Βάδη Βιρτεμβέργη, μπορείτε να δείτε και το βιντεάκι στο YouTube, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Αρχικά, λοιπόν, να σας πω πως το νομικό πλαίσιο δεν είναι ε, νομικό πλαίσιο, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά αυτά που λύνει. Αυτό οφείλεται στον ε, κανονισμό για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Έχει διάφορες ονομασίες, ε, δεν υπάρχει σωστή οργάνωση. Από τη μία τον ονομάζουμε ΕΣΥ, κανονισμό ΕΣΥ, ESIF, CSF, έχει διάφορες ονομασίες. Μετά, από την άλλη, υπάρχει και ο κανονισμός για τα περιφερειακά ταμεία. Τέσσερι, ε, εφτά εφαρμοστικές διατάξεις, τρεις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, μία διορθωτική. Υπάρχει λοιπόν ένα σωρός, ένα συνονθήλευμα διαφορετικών ε, κανονισμών, το οποίο έχει οδηγήσει στο να υπάρχει τέτοια σύγχυση που να ξεχάσουν οι διοικητικές αρχές ποιος είναι ο κανονισμός που πρέπει να εφαρμόσουν. Περνάω τώρα στο επόμενο σημείο της παρουσίασής μου. Θεωρώ πως ε, το ταμείο, τα περιφερειακά ταμεία και το Ταμείο ε, Γεωργικής Ανάπτυξης της Υπέθρου είναι τελείως ασύμβατα. Αυτό εδώ είναι το ε, περιφερειακό, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 17 άρθρα, 13 ενίες. Αυτό εδώ είναι το Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης, 90 άρθρα, 62 σελίδες. Βλέπουμε λοιπόν ότι η νομοθεσία είναι τελείως διαφορετική και ε, τελείως διαφορετικά τα σημεία στα οποία εστιάζει. Έπειτα, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, υπόκειται στην ε, εξουσία των ε, των, ε, χωρών, των επιδοτήσεων. Υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικές λοιπόν νομοθεσίες. Μετά, να σας ε, ενημερώσω και για κάποιες επιπλέον διαφορές υπάρχουν οι διαφορές στις λεγόμενες μικρές ε, υποδομές, μικρά έργα υποδομών. Η συνάδελφος ήδη το ανάφερε. Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Ταμείο και στο Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης της Υπέθρου συνυπολογίζονται στα καθαρά έσοδα. Είναι το απλοποιημένο κόστος, simplified cost. Και αυτά ε, χρησιμοποιούνται και για τον ε, λογιστικό έλεγχο. Τι είναι λοιπόν αυτές οι μικρές υποδομές. Στα πλαίσια του Ταμείου Γεωργικής ανάπτυξη είναι διάφορες, ε, διάφορα μικρά έργα, διάφορα, σήμανση μονοπατιών, διαδρομών κτλ. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ορίσει το ίδιο ποιο θα είναι το ύψος ε, των ε, δαπανών. Σε εμάς ανέρχεται στα 600.000 ευρώ, από 30 μέχρι 600.000 ευρώ. Πολύ μεγάλο ευρώς. Μετά, το κόστος ε, ανεβαίνει όταν πάμε σε περιπτώσεις ε, μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς, όπου εκεί μπορούν να διτεθούν ε, το πολύ 5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν μετά διάφορες ομάδες, διάφοροι διαχειριστικοί φορείς, οι οποίοι αποφασίζουν για το ύψος των επιχορηγήσεων. Όμως, δεν έχουν καμία οικονομική ευθύνη. Διαφορετικά όμως είναι τα πράγματα για τις ε, δημόσιες αρχές. Στο Περιφερειακό Ταμείο οι δημόσιες αρχές είναι οι μόνες οι οποίες έχουν αρμοδιότητα για την επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με το, ε, το άλλο ταμείο. Πρέπει να έχουν γραπτεί η άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να διεξαχθεί μια μελέτη εκτύπου, να δούνε αν όλα είναι σωστά, αν, υπάρχουν, αν έχουν γίνει σωστές, ληφθεί σωστές αποφάσεις, αν έχουν γίνει σωστές μελέτες, αν υπάρχει σωστή κατάρτιση του προσωπικού, αν, υπάρχει, αν υπάρχουν κανόνες για την, για την πρόληψη της απάτης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι ε, η εποπτεία είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όποιος αναλαμβάνει την εποπτεία το κάνει με δική του ευθύνη και καλά να πάθει. Τώρα, περνάμε στα καθαρά έσοδα. Στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο άρθρο 65, τα καθαρά έσοδα, για παράδειγμα για διάφορα ενευνητικά προγράμματα, ε, ανήκουν στις, ε, στις, ε, στο διοικητικό φορέα, στον ορίζοντα 2000 οι 20 όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το ε, κόστος πηγαίνει στο, στο ερευνητικό ε, ίδρυμα, όμως αυτό περιπλέκει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Να σας αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα για τα καθαρά έσοδα. Το 2014 θεωρήθηκε ότι η εξοικονόμηση πόρων θεωρείται και αυτή ε, καθαρό έσοδο. Ας δούμε την περίπτωση ενός παιδικού σταθμού, βρεφονοπιακού σταθμού, κάτι που είναι συνηθισμένο φαινόμενο στη Γερμανία. Αν α πούμε ανέβει η τιμή του πετρελαίου θέρμανση σε έναν κρύο χειμώνα, τότε θα ε, πρέπει να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα για θέρμανση, γιατί τα παιδιά πρέπει να έρχονται σε ένα καλά συσταμένο χώρο. Στον επόμενο χειμώνα όμως, αν δεν είναι τόσο κρύος, ε, τότε αλλάζουν τα δεδομένα και εκεί υπάρχει περιθώριο λάθους. Περνάμε τώρα στο απλοποιημένο κόστος. Είναι κάτι που αγαπώ ιδιαίτερα, όπως θα δείτε. Κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές, 60 ολόκληρες σελίδες για το απλοποιημένο κόστος, γεμάτες μπλα μπλα, γεμάτες πολυγίες, τις οποίες πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε. Και τα κράτη μέλη έχουν ε, την ε, δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις και οι ερωτήσεις αυτές που ε, ετέθησαν καλύπτουν 35 σελίδες για, τα, για το απλοποιημένο κόστος. Εάν βρείτε απάντηση, εγώ θα φάω τη γιαγιά μου. Ας περάσουμε τώρα και στα χρηματοδοτικά μέσα. Είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση, είναι αρκετά πολιτική. Δεν θα ήθελα λοιπόν να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα σας αναφέρω ενδεικτικά ότι υπάρχουν 30 διαφορετικές αρμόδιες αρχές και είναι αναπόφευκτο να συμβούν λάθη. Τα χρηματοδοτικά μέσα λοιπόν τα βλέπετε εδώ. Κρατάω αυτό το πανάλαφρο πακέτο 2,5 κιλών. Αυτά λοιπόν είναι τα χρηματοδοτικά μέσα και πρέπει να τα γνωρίζουμε όλα. Αυτοί λοιπόν οι κανόνες είναι η αιτία που δημιουργούνται λάθη. Αλλά ας περάσω τώρα στα λογιστικά. Είναι το καλύτερο κομμάτι της παρουσίασής μου. Όπως ξέρετε, υπάρχουν διάφορες αγροτικές επιδοτήσεις. Εκεί ο αγρότης ε, λαμβάνει ε, ε, επιδοτήσεις ανάλογα με, το, με την έκταση της εκμετάλλευσής του. Όταν τελειώνει λοιπόν το οικονομικό έτος, τότε γίνονται και οι λογαριασμοί. Εάν στο τέλος παρατηρήσω ότι μετά από επιχορηγήσεις για ένα έργο που καλύπτει έξι χρόνια δεν φτάνουν ή δεν έχει γίνει κάποιος, κάποιος λάθος υπολογισμός, τότε πρέπει όλο αυτό το ποσό να επιστραφεί και η γραφειοκρατία που δημιουργείται είναι απίστευτη. Έπειτα, οικονομικό έτος. Δεύτερο σημείο που αξίζει να σας ε, αναφέρω. Πληρω... Οι πληρωμές κατα... γίνεται... Ε, πληρωμές καταβάλλονται μετά τον ε, ισολογισμό του οικονομικού έτους. Όμως, κάθε έργο, το οποίο αποτελείται από διαφορετικά επιμέρους έργα, έχει και διαφορετικούς λογαριασμούς και διαφορετικές δαπάνες. Έχουμε λοιπόν εκατοντάδες αποδείξεις, οι οποίες πρέπει κάθε μία από αυτές εξεχωριστά να μπορούν να ε, εξεταστούν για να δούμε εάν έχουν γίνει σωστά, εάν έχει γίνει κάποιο λάθος. Αυτό μάλιστα πρέπει να συμβαίνει σε βάθος ε, όλων των ετών που διαρκεί ένα πρόγραμμα. Αυτό δημιουργεί μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος και χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε μία λύση που θα είναι προσανατολισμένη σε αποτελέσματα και σε λύσεις και όχι να τα δημιουργεί όπως τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποια πορίσματα από αυτά τα οποία ακούσαμε και ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα παραδείγματα τα οποία παρουσιάστε. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον καθηγητή Βασίλε Ντουκάρο από το Πανεπιστήμιο της Τιμισουάρα στην Ρουμανία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας πρώτα απ' όλα. Τα η παρουσίασή μου βασίζεται στην εμπειρία μου. Έχω τέσσερα χρόνια δραστηριότητα σε ένα ενδιάμεσο οργανισμό, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα και την καινοτομία, την τεχνική διαδικασία συντονισμού μέσα στο Πανεπιστήμιο για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι απόλυτες στρατηγικές σε επίπεδο νουτς 3 στην περιοχή της Τιμισουάρα ώστε να υπάρξει καλύτερη περιφερειακή ανάπτυξη. Έχουμε δει την έκθεση του κυρίου Τσεντρόνε του Ιουνίου του 2011 από το Ελεκτικό Συνέδριο. Θα ήθελα λοιπόν να πω καταρχήν ότι θέλω να ευχαριστήσω τον Δόκτωρ Αρίς για την συνεργασία μου, για να με βοηθήσει στην παρουσίασή μου. Και είναι φανερό ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι στόχοι προτεραιότητος, κάποιες ε, αξιολογήσεις και να υπάρχουν κοινοί ενδείκτες στο έργο μας. Επίσης αναφερόμαστε στην απλοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης. Και αυτό μας ενδιαφέρει σήμερα γενικά είναι η απλοποίηση των διαδικασιών γιατί είναι φανερόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε ότι αφορά την χρήση των ευρωπαϊκών μέσων, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πραγματικά ευφύης εξειδίκευση στα θέματα αυτά για να επιτευχθεί η απαραίτητη αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την χρησιμοποίηση των πόρων και επίσης να υπάρχει μια αντίστοιχη αποδοτικότητα στην διαδικασία αξιολόγησης της χρήσης αυτών των πόρων. Για ένα Ινστιτούτο στη Σεβίλη ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή και έχουν προσπαθήσει να μετρούν τις διάφορες ροές μεταξύ περιφερειών. Ο στόχος είναι να καταμετρηθούν οι διάφορες χρηματικές ροές και με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούσαν, θα μπορούσαν να καταμετρήσουν μια σημαντική οικονομική ε, μεταβλητή που είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα. Όταν λοιπόν θέλουμε να πετύχουμε ε, την απλοποίηση θα πρέπει να σκεφτούμε για, σε διάφορους τομείς. Από τη μια μεριά είναι η επιστημονική γνώση, από την άλλη μεριά είναι το δίκαιο το οποίο διέπει τα θέματα αυτά και το τρίτον είναι οι εμπειρικές διαδικασίες. Για τα νομικά θέματα μίλησε ήδη ο προηγούμενος ομιλητής για τα, εμπορικά, για τα εμπειρικά θέματα μας ενδιαφέρει να έχουμε τις σωστές μετρήσεις. και επίσης μας ενδιαφέρει να έχουμε λιγότερη συλλογή δεδομένων, αλλά έχουμε πιο ουσιαστικά δεδομένα. Αυτό θα είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της απλοποίησης όπως τη βλέπουμε, δηλαδή να υπάρξει λεγόμενη ευφυής εξειδίκευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπροστά της πολύ θετικά αποτελέσματα, πολύ καλές εμπειρίες από την έρευνα και την ανάπτυξη και τα προγράμματα καινοτομίας το, υπάρχει το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Χρόνιγεν, όπου έχουν ε, γίνει προσπάθειες να εκτιμηθούν οι ροές προστιθέμενης αξίας στις συναλλαγές μεταξύ κρατών. Και έχει γίνει αυτή η καταμέτρηση σε επίπεδο σορευτικό, σε επίπεδο των περιφερειών του, της κατηγορίας νουτς 2. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνει αυτή η καταμέτρηση σε διάφορα επίπεδα ώστε να μπορούμε να επιτύχουμε την σύγκληση και την συνοχή σε οικονομικό επίπεδο και επίσης και ένα βαθμό εξειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί απόντος της εξειδίκευσης αυτής δεν θα μπορέσουμε παρά να καταλήξουμε στο να χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα για να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα σε δύο, τρεις και περισσότερες περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κυρίως πώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιαστούν ώστε κατά τη διαδικασία της παραγωγής θα χρησιμοποιούνται λιγότεροι φυσικοί πόροι και ενέργειες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εξειδίκευση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν καταλαβαίνουμε πώς, ε, ποιο είναι το περιεχόμενο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Εμείς πρέπει να βασιστούμε σε ένα αριθμό βασικών ενδεικτών με στόχο να αναπτύξουμε ορισμένες ε, δράσεις. Μας ενδιαφέρει να καταμετρήσουμε καταρχήν την ε, παραγωγικότητα ορισμένων τομέων. Παραδείγματος χάρη αν πάρουμε την Αυστρία. Στην Αυστρία ως παράδειγμα είχαμε προτείνει να κατηγορηποιήσουμε τους τομείς επί τη βάση της εξειδίκευσής τους όπως γίνεται και για τα θέματα έρευνας. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να καταλάβουμε Πώ αυτέ οι εταιρικέ σχέσει θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Γιατί χωρί αυτέ τι εταιρικέ σχέσει είναι αδύνατο να φτάσουμε σε επίπεδο εξειδίκευση. Θέλουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό τη εξειδίκευση, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε συνεχτικές και σταθερέ προσπάθειε. Έχουν δημοσιευτεί κάποια στοιχεία για το 2011, τα οποία μας δίνουν δυνατότητα με αυτή την απογραφή να ξέρουμε πόσες είναι οι, εργατικές, οι εργασόμενοι στο στην εργασιακή δύναμη και πρόκειται για μια μελέτη η οποία αφορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε κατατάξει όλους τους εργαζομένους επί τη βάση της ηλικία τους, του εργασιακού κλάδου, της φυλής τους. Είχαν καταμετρηθεί όλα αυτά λοιπόν. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση η εμπειρία των Γερμανών μελετητών έχει οδηγήσει σε μια νέα διαδικασία καταμέτρησης των υλικών και των υπηρεσιών σε μακροοικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένων προϊόντων. Θα πρέπει λοιπόν να το κάνουμε αυτό ώστε να μπορούμε να καταμετρήσουμε την προσθέμενη αξία και να δούμε κατά πόσο είναι λυσιτελής η χρήση των φυσικών Είναι απαραίτητο λοιπόν τα συστήματα αυτά με τους ενδείκτες να χρησιμοποιηθούν και με τον τρόπο αυτό στο χαμηλότερο επίπεδο, στο νουτς 3, να χρησιμοποιηθούν και φυσικά να σωρευτούν μέχρι του επίπεδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί βλέπουμε ότι οι καταμετρήσεις στους διάφορες περιοχές γίνονται με διαφορετικό τρόπο και δεν είναι ομοιογενείς. <coughs> Σημαντικό λοιπόν οι εταιρικές σχέσεις να μην γίνονται μόνο μεταξύ δύο περιοχών, αλλά μεταξύ και περισσότερων και να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συνεργασίες ερευνητικών ομάδων. Αλλιώς κινδυνεύουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια να χρησιμοποιούνται δύο και τρεις φορές για τον ίδιο σκοπό. Οι μεταφορές λοιπόν κονδυλίων θα πρέπει να βασίζονται και στις μεταφορές τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειών έχουμε μιλήσει για τη λεγόμενη αποσύνδεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να έχουμε αποσύνδεση της παραγωγής στο βαθμό του δυνατού από τους φυσικούς πόρους και την ενέργεια, ενώ συγχρόνως αυξάνουμε την παραγωγικότητα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, μια εξειδίκευση αφενός, αλλά και μια σταδιακή αποσύνδεση από, τους πρώτους, από τις πρώτες ύλες και την ενέργεια που θα μας οδηγήσει σε σημαντικές εξα, εξοικονομήσεις για την αποσύνδεση αυτή όπως είπαμε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει υπό η υποστέμενη αξία. Δηλαδή δεν θα υπάρξει απώλεια προστέμενης αξία. Μίλησα λοιπόν για αυτού του τρει στόχου. Καταρχήν να υπάρξει σύγκληση και συνοχή και μετά στο δεύτερο χρόνο να περάσουμε σε μια ευφυή εξειδίκευση. Έχουμε λοιπόν αυτές τις ε, μερικές εμπειρίες, αλλά θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε ακόμα πιο εξελιγμένα και κοφτερά εργαλεία για να μπορέσουμε να έχουμε τους απαραίτητους δείκτες με τους οποίους θα είναι στη συνέχεια πιο εύκολο να έχουμε τη σωστή μέτρηση της ε, χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων και υπάρχει μια μελέτη από το Ινστιτούτο της ε, Σεβίλης για τα θέματα αυτά πώς μπορεί κανείς να καταμετρήσει τις εμπορικές ροές μεταξύ περιφερειών της ε, Ευρώπης και υπήρξε μια μελέτη για την περιοχή του Βερολίνου το 2010. Και προέκυψε λοιπόν από τη μελέτη αυτή μία σειρά από προτάσεις για μέτρα ώστε να υπάρξει ε, καταμέτρηση της χρήσης πόρων και ενέργειας και επομένως πώς συνδέεται αυτό με την προσθέμενη αξία και επίσης στο Πανεπιστήμιο του Κρόνιγκεν έχουν γίνει ε, μετρήσεις εμπορικών ροών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κίνα και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και ίσως μπήκα σε κάποιες λεπτομέρειε εδώ μιλώντας για τα, το θέμα του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν έχουμε 28 κράτη-μέλη μπορούμε να προωθήσουμε μία εξειδίκευση των χωρών αυτών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ή τους τομείς παροχής υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό όλες αυτές οι χώρες θα επωφεληθούν. Θα είναι αυτό λοιπόν μια πολύ σημαντική πρόκληση. Όπως είχε πει ο μακαρί της νομπελίστας κ. Σάμουλσον τη δεκαετία του 70. Και θα μας οδηγήσει λοιπόν σε μια καλύτερη χρήση των ε, διαφορετικών πόρων από τις επιχειρήσεις και συνολικά θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό συμφέρον μεταξύ επιχειρήσεων και τοπικών και περιφερειακών αρχών. Και έτσι, από τη μια μεριά θα εξασφαλίσουμε την κερδοφορία που επιδιώκουν οι επιχειρήσεις, αλλά συγχρόνως θα προωθήσουμε και το κοινό συμφέρον που επιθυμούν οι Δήμοι και οι τοπικές αρχές. Και θα έχουμε και την σωστή ε, νομοθετική ρύθμιση. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα της, στην περίπτωση της Αυστρίας. Βλέπουμε τι έχει επιτύχει η Αυστρία σε επίπεδο Εξειδίκευση. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν τομείς όπου υπάρχει δημιουργία προσθέμενης αξίας αλλά με έμεσο τρόπο. Μπορούμε από αυτό να βγάλουμε το εξή συμπέρασμα. Η Αυστρία είναι από τις λίγες χώρες που σε επίπεδο χώρας έχουν καταφέρει να, να ακολουθήσουν αυτήν την οδό της εφιούς Δηλαδή μέτρησαν τις εισρωές και εκροές της παραγωγής και την προσθέμενη αξία σε κάθε περίπτωση. Έτσι μπόρεσαν να παρακολουθήσουν στοιχεία όπως παραγωγός η παραγωγικότητα σε διαφορε τομεί, η αντίστοιχη κίνηση των αποδοχών των εργαζομένων. Έχουμε λοιπόν αυτό το εργαλείο το οποίο έχει δημιουργηθεί και αυτό έχει γίνει ε, με τη βοήθεια της Eurostat με την αίτηση της Eurostat, αν θέλετε καλύτερα, μια ομάδα από Γερμανούς ερευνητές της Χαϊδερβέργης, του Αμβούργου και άλλων πανεπιστημίων προχώρησε σε μια συγκεκριμένη μέτρηση που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Το σημαντικό είναι ότι, θα γίνει αυτή, ότι πρέπει να γίνει αυτή η καταμέτρηση σε λεπτομεριακό επίπεδο. Φυσικά πρέπει να συμπεριληφθούν και τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης των ε, ε, απορριμμάτων κτλ. Και εδώ έχω αναφέρει ένα παράδειγμα σε επίπεδο κατανάλωσης που έχει να κάνει με διάφορες μορφές κατανάλωσης ε, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι βλέπουμε λοιπόν. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει μειωθεί μόνο λίγο αυτή η κατανάλωση πόρων και η ανακύκλωση είναι περιορισμένη. Τέτοιους δείκτες θα πρέπει να καταμετρούμε σε όλα τα σχέδια ώστε να μπορούμε να βλέπουμε κατά πόσο προχωρούμε προς το στόχο αυτό που επιδιώκουμε, που πρέπει να επιδιώκουμε και τον οποίο τον ονόμασα ευφυά εξειδίκευση. Όλα αυτά λοιπόν με οδηγούν να παραπέμψω και στην μελέτη αυτή που έγινε από το που ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την χρήση των φυσικών πόρων. μια ομάδα Γερμανών ε, ερευνητών, περίπου 100, που έκανε αυτή τη μελέτη και μετά υπήρξε μια παρέκβαση αυτών των στοιχείων και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία υπολογισμού ε, στοιχείων που εμείς έχουμε αντλήσει από την περιοχή του Τίμης, δηλαδή στην ε, ενδοχώρα της Τίμης Οάρα στην ε, Ρουμανία, σε σχέση με τη χρήση πόρων και σε σχέση με την εξέλιξη της ε, παραγωγικότητος και την ε, δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Ε, σε επίπεδο περιοχής είναι δύσκολο βέβαια να δει κανείς αν πράγματι επιτυγχάνεται αυτή η ευθύης εξειδίκευση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο λεπτομερείς μελέτες και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνεται με πιο απλό τρόπο αυτή η διαδικασία καταμέτρησης και ίσως να σας κάνω τώρα μία σύνοψη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς μία ευφυά εξειδίκευση η οποία θα βασίζεται στην έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος να καταμετρήσουμε την χρήση φυσικών πόρων και την χρήση ενεργείας και να βασιστούμε φυσικά στις ε, ευρωπα... ευρωπαϊκές στατιστικές της Eurostat αλλά και στις εθνικές ε, στατιστικές και μετά θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να λειτουργήσει αυτή η εξειδίκευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία τα οποία είναι τόσο εύκολα να χρησιμοποιήσει κανείς και μπορούν να μας επιτρέψουν να έχουμε μια συσσόρευση στοιχείων σε διάφορα επίπεδα και σε χώρες όπως η Ρουμανία παραγματικά χάρη υπάρχει ένα παράδοξο στον εργασιακό χώρο. Μέχρι το 2020 θα μειωθεί ο πληθυσμός μας, θα χάσουμε περίπου ένα εκατομμύριο ε, ανθρώπων οι οποίοι δεν θα μπορούν. Θα χρειαστούμε δηλαδή να βρούμε ένα εκατομμύριο ανθρώπους που θα εργάζονται για να μπορέσουμε να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα παραγωγής. Συζητάμε πάρα πολλέ φορέ λοιπόν για κανόνε και στρατηγικέ. Πρέπει να είναι ολοκληρωμένε, όμω αυτέ οι στρατηγικέ θα πρέπει να εφαρμοστούν σε συνολικό επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα, πάρα πολλέ στρατηγικέ που δεν είναι συνδεδεμένε μεταξύ του. Το είπε και ο προλαλή σα μου. Είναι μεμονωμένε πολλέ φορέ αυτέ οι στρατηγικέ. Προσπάθησα λοιπόν με όλα αυτά που σα είπα να εξηγήσω τι σημαίνει αυτή η εξειδίκευση, αυτή η ίδια η εξειδίκευση έχει μεγάλη σημασία στην Ρουμανία, παραδείγματο. Χάνονται πάνω από 5 δισεκατομμύρια, εκτιμάται, από την έλλειψη ε, εξειδικευσής. Αυτή λοιπόν η κοινή μέθοδος καταμέτρησης η οποία παρουσιάστηκε εδώ και η οποία οδηγεί στην αποτελεσματική χρήση των πόρων και της ενέργειας είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εφαρμόσουμε. Δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μονάχα στο σεβασμό των κανόνων, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν σπαταλώνται και οι πόροι. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να καταλήξουμε σε ένα υπόδειγμα σε ό,τι αφορά την εργασιακή δύναμη. Αλλιώ δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την εξειδίκευση τη εργασιακής δύναμη και ε, παράλληλα θα πηγαίνει χέρι με χέρι αυτή η στρατηγική με την στρατηγική για την χρησιμοποίηση σε αποδοτικό επίπεδο των φυσικών πόρων και φυσικά με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη υποστήριξη στους νεοφανείς τομείς της οικονομίας ώστε να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την μεγέθυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την κάπως διαφορετική προσέγγιση που παρουσιάσατε επί του θέματος της απλούστευσης. Συνάδελφοι, έχετε το λόγο. Ερωτήσεις, ερωτήσεις, προτάσεις, κύριε Νοβάκοφ κύριε Έθεριτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που έχουμε εδώ δικαιούχους και το εκπροσώπους των τοπικών αρχών για να συζητήσουμε τις πολιτικές συνοχές, γιατί οι πολιτικές συνοχές αφορούν τους πραγματικούς πολίτες, όχι τους εργαζόμενους στα ευρωπαϊκά όργανα. Οπότε αυτή η δικαιούχοι, αυτοί οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών είναι στην πραγματικότητα ε, το ραντάρ σε ένα αεροδρόμιο που λέει στο αεροπλάνο που να πάει. Δεξιά αριστερά, πάνω κάτω. Ξέρετε, μερικές φορές εμείς ζούμε μέσα σε ένα παραμύθι. Πιστεύουμε όλοι ότι όλα πάνε καλά, αφού ψηφίσαμε εμείς υπέρ και θεωρούμε ότι όλα πάνε μια χαρά. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Μπορούμε να συζητάμε ε, επί ώρες για τα προβλήματα και λέτε εσείς κυρίες ότι είναι πολύ χαρτούρα να πού να δείτε τι έχουμε εμείς ε, στο πρόγραμμα μέχρι το 2020. Μπορούμε να μιλήσουμε βεβαίως και να επεκταθούμε πολύ ε, για τα προβλήματα, αλλά καλό θα ήταν να μιλήσουμε και για κάποιες λύσεις. Η γραφειοκρατία και τα ο διοικητικός φόρτος ενίοτε αποθαρρύνουν τους δικαιούχου από το να συμμετάσχουν στην ε, πολιτική συνοχή. Την ε, αποφεύγουν ουσιαστικά. Μάλιστα μερικέ τοπικέ αρχές και κάποιες εταιρείε ε, προτιμούν να πάρουν δάνειο από τράπεζα και να το εξοφλήσουν μετά αντί να περάσουν από τις κοινοτενείς απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε το 8% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στα, τα διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη και οι τοπικές αρχές. Είναι η βασική κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας και δεν μπορούμε εμείς να θέτουμε τόσα εμπόδια σε αυτούς τους δικαιούχους. Αφού συζητήσαμε λοιπόν για τόσα προβλήματα, εγώ θα ήθελα να κάνω μερικές προτάσεις και να ακούσω τις απόψεις των καλεσμένων μας. Πιστεύω ότι αν είχαμε παρόμοιες ή τουλάχιστον τυποποιημένες διαδικασίες ε, δημοσίων συμβάσεων, ε, τα πράγματα θα ήταν ευκολότερα. Φανταστείτε ότι εγώ έχω μια επιχείρηση και με ενδιαφέρουν οι δημόσιε συμβάσει στι κατοχώρε και στην Πολωνία. Δύο εντελώ διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια, δύο εντελώ διαφορετικέ διαδικασίε και αυτό με κάνει, με διώχνει ουσιαστικά αντί να πάω σε αυτέ τι χώρε. Ποια θα μπορούσε να ήταν η λύση. Γιατί να μην απλουστεύσουμε τις διαδικασίες ελέγχου. Πώς θα ήταν αν ο έλεγχος ε, όλων των θεσμών ήταν παρόμοιος. Ε, μπορούσε να γίνει από κοινού από όλους τους θεσμούς, αντί να ε, ελέγχουμε το ίδιο πρόγραμμα δύο ή τρεις φορές. Αυτή ήταν μια ιδέα που είχα. Θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη των συναδέλφων και των προσκεκλημένων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ο κ. Σέφερετς να σας ζητήσω να ε, είστε σύντομοι ώστε να υπάρξει χρόνος για απαντήσεις. Έχουμε περάσει πάνω από μια ώρα ακούγοντας την αρπαστικές ομιλίες υπέρ της απλούστευσης και τα συγχαρητήριά μου προς ομιλητές. Είναι σαν να βρίσκομαι με ακαδημαϊκές διάνοιες ε, μέσα στην αίθουσα αυτή, πανέξυπνοι, ευφύς άνθρωποι, πολύ καλοί. Αλλά ξέρετε, δεν είναι αυτή η απλούστευση που θα ανέμενε ο καθής. Από όσο κατάλαβα ως απλός άνθρωπος, εσείς μιλήσατε για απλούς τρόπους για να επιτευχθούν περισσότερα. Απλούς τρόπους για να δαπανηθούν περισσότερα, να φέρουμε περισσότερα αποτελέσματα. Ενώ πολλές φορές ε, σε αυτή την επιτροπή λέμε ότι τόσο δεν υπάρχουν τα λεφτά για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, η πραγματική απλούστευση θα μπορούσε να βασιστεί σε έναν πιο σαφή ορισμό του πώς μπορούμε να κάνουμε λιγότερα μεν, αλλά πιο αποτελεσματικά και πιο απλά. Μεγάλο κομμάτι της συζήτησης σήμερα αφορούσε το πώς να κάνουμε περισσότερα, αλλά πιο αποτελεσματικό για τους γραφειοκράτες. Και η ερώτηση με εμένα ως απλό ανθρώπου είναι, έχει περάσει από κανενός το νου ότι όλες αυτές οι σκέψεις, όλη αυτή η ευφυΐα που επενδύεται σε αυτό το τεράστιο ακαδημαϊκό και γραφειοκρατικό μηχάνημα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερο αν κάναμε λιγότερα με καλύτερο τρόπο και με πιο δημοκρατικό τρόπο δηλαδή να ε, ε, δώσουμε αποτελέσματα που να ικανοποιήσουν περισσότερους ανθρώπους. Ε, ευχαριστώ βέβαια όλους τους ακαδημικούς που βρέθηκαν εδώ και για τις εξαιρετικές τους ομιλίες και για όλες τις πληροφορίες. Κυρία Βάνεκ, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και όλους τους εμπειρογνώμονες για αυτές τις εξαιρετικές παρουσιάσεις και για τις συγκεκριμένες προτάσεις που μας έκαναν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας να διεξάγουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με τέτοια μυαλά έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα. Πιστεύω πως η απλούστευση της γραφειοκρατίας είναι πολυδιάστατη. Υπάρχει από τη μία η διάσταση της διαφάνειας, δηλαδή λήψη αποφάσεων σχετικά με την απλούστευση, αντικειμενικές ε, διεξαγωγές ανάλυσης, αξιολογήσεις. Υπάρχει από την άλλη η δημοκρατική, ε, η πολιτική άποψη, δηλαδή τη σχέση έχω εγώ, πώς με αφορά εμένα αυτή η απλούστευση και ε, επίσης υπάρχει και η άποψη της αναλογικότητας που μας απασχολεί εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι γίνεται με τις ε, επιχειρήσει, επιχειρήσεις, πώ επηρεάζει εκείνε, αλλά επίση και μια ποιοτική άποψη, δηλαδή πώ ποιοτικά μπορώ εγώ να επιτύχω του στόχου της Ευρώπη 2020, Πώ μπορώ να συνεισφέρω, να βάλω και εγώ το δικό μου μικρό λιθαράκι για αυτόν τον στόχο. Για παράδειγμα, πώ θα δώσουμε κίνητρα για διάφορα ε, βιώσιμα έργα, αηφόρα έργα και αυτή είναι και η πρώτη μου ερώτηση. Εσεί ε, τι ε, πρόταση έχετε για την απλούστευση της ε, ποιότητας. Και μία ερώτηση στον ε, κύριο Ρης. Μας είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτά τα δύο ταμεία, πως δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Μπορείτε να μου δώσετε περισσότερες ε, πληροφορίες, δηλαδή να μας πείτε κατά την άποψή σας ποια είναι, ε, ποιοι είναι οι λόγοι, ποια είναι τα προβλήματα και, ε, που μπαίνουν εμπόδιο στην προσέγγιση αυτών των δύο ταμείων και τι προτείνετε εσείς να γίνει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Όλμπριχτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω πως αυτή η συζήτηση έχει πολλές στοιχείες. Μία είναι η δομή της πολιτικής συνοχής. Και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για τις σχέσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πολιτικές, είναι στη σχέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στις σχέσεις μεταξύ των διαφορών γενικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμα και για τις σχέσεις μεταξύ των διαφορών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμα και για τη σχέση μεταξύ των διαφορών πολιτικών ομάδων εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελείω διαφορετικέ προσεγγίσεις όχι μόνο από τι πολιτικέ ομάδε, αλλά και από τι επιτροπέ. και εδώ δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε μεταξύ μα γιατί ο καθένα πολεμά για τα δικά του συμφέροντα. Έχουμε ας πούμε τους, ε, τα μέλη της Επιτροπής ε, Απασχόλησης που προσπαθούν να επερασπιστούν τα δικά του συμφέροντα έναντι της, πολιτικής, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ξέρετε πολύ καλά πώς είναι αυτά τα πράγματα. Δημιουργείται μια σύγχυση, ένα κουβάρι από το οποίο προσπαθεί ο καθένας να κερδίσει τα περισσότερα. Και δεν ξέρω εάν η ενοποίηση είναι ε, κατάλληλη, αν ε, μήπως χρειάζεται να υπάρχουν ξεχωριστά τα μία ξεχωριστές λύσεις. Εγώ πιστεύω πως η λύση που προτείνατε εσείς, το ένα κοινό ταμείο είναι η πιο τίμια. Είναι μια λύση που δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, μια ξεκάθαρη προοπτική. Μας λέει φτάνει πια. Φτάνει πια αυτό το χάλι, πολιτικά και οικονομικά. Ένα λοιπόν κοινό ταμείο, μία κοινή πολιτική, ένα κοινό οδικό χάρτη. χάρτης. Διαφορετικά αυτή η διαδικασία απλούστευση θα καταλήξει να μπερδέψει περισσότερο το κουβάρι και μετά θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε μια άλλη διαδικασία όπου θα εξηγούμε πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η διαδικασία απλούστευσης. Δεν θα επεκταθώ, καταλαβαίνετε πιστεύω ότι εννοώ, αλλά αυτά είναι απλά δημοσιονομικά. Και την περασμένη εβδομάδα νομίζω πάλι είχαμε μια παρόμοια συζήτηση για τους ε, δείκτες ε, στην, στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Ελάχιστοι πιστεύουν πως το θέμα είναι το πώς να διεξάγει σωστά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Οι περισσότεροι θέλουν να ελέγχουν τον προϋπολογισμό, θέλουν την, την εξουσία. Και φυσικά ξέρετε ότι το τίμημα για αυτόν τον έλεγχο είναι μεγαλύτερο από το κέρδος που ε, αποκομίζουμε από τα διάφορα έργα. Αυτό οδηγεί και στην ε, μείωση του ενθουσιασμού, σε λιγότερα κίνητρα για να αρχίσουν έργα και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Φυσικά αυτά τα κίνητρα είναι ξεκάθαρα. Χρειάζονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Λιγότερο από τα διαρθρωτικά ταμεία και εάν αυτά τα κονδύλια δεν είναι αρκετά τότε υπάρχει μια, αυτή, μια τάση παρέτησης. Γι' αυτό λοιπόν αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία βλέπουμε ότι η πολιτική ηγεσία σιγά σιγά θα κατανοήσει το όφελος, θα πει ευχαριστώ, είναι προς το όφελος των πολιτών μας. Όμως ε, στα υπόλοιπα, στα πιο μικρά κράτη θα πούν ότι δεν αξίζει τον κόπο, είναι λιγότερα ε, τα κονδύλια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σκεφτείτε ότι λιγότερα κονδύλια με περισσότερη γραφειοκρατία οδηγούν σε απογοήτευση, οδηγούν στο, το, τους... Ε, πολίτες να αναζητούν χρηματοδότηση αλλού. Ένα λοιπόν κοινό ταμείο. Αυτό είναι η λύση. Και να μην εστιάζουμε στον έλεγχο αλλά στο, στον τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φανής έχει το λόγο. Θα ήθελα να σχολιάσω τις ε, παρεμβάσεις που ακούσαμε σήμερα που ήταν πολύ καλές. Αυτό το οποίο θα ήθελα το, το θέμα της μεταρρύθμισης της, ε, των δημοσιονομικών προοπτικών για το οποίο θα είναι ο η ε, εισηγητής. Θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι απόψεις στο σημείο αυτό. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα ψήφισμα εξ ονόματος του Κοινοβουλίου σε λίγες μέρες από τώρα Οπότε μας δώσετε μερικές βασικές ιδέες που θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στη συζήτηση. Thank you. Thank you. Madame Bresso. Η κυρία Μπρέσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Και εγώ με την εμπειρία που έχω στον τομέα συμφωνώ με τα όσα είπε ο συναδελφός κύριος Σόλμπερτ. Όταν μιλάμε για απλούστευση, αυτό μεταφράζεται σε δύο πτυχές. Πρώτα απ' όλα τη διαφορά των κανόνων μεταξύ των διαφορετικών ταμείων που εμποδίζουν την πολυ, τον πολυταμιακό προγραμματισμό που είναι ένας από τους προηγμένους στόχους της νέας προγραμματικής περίοδου. Οπότε γι' αυτό πρέπει να είμαστε ε, αμετακίνητοι την επόμενη φορά θα πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ως Επιτροπή για να συμφωνήσουν και οι Επίτροποι μεταξύ τους Υπάρχουν ναι, ναι, διαφορετικές πολιτικές, αλλά τα διάφορα ταμεία πρέπει να έχουν τους ίδιους κανόνες για να μπορέσει να υπάρξει πολυταμιακός προγραμματισμός. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι ναι, να δίνουμε τεράστια προσοχή στα αποτελέσματα, αλλά δεν μπορούμε για να το κάνουμε αυτό να διατηρούμε τους ίδιους κανόνες. Θα πρέπει να ελαφρύνουμε τους επίσημους ελέγχους και τους οικονομικούς ελέγχους πέραν του τελευταίου που αφορά τη συμφωνία μεταξύ του κόστους και του αποτελέσματος γιατί αλλιώς ο κίνδυνος ε, κατά το επαλήθευση του αποτελέσματος ε, θα επιδεινώνεται λόγω των περαιτέρω γραφειοκρατικών ε, επιπλοκών. Ειδικότερα σε περιπτώσεις όπως σαν οι συναδέλφοι όπου οι επενδύσεις είναι μικρές σχετικά απλά για την ενεργοποίηση ε, προγραμμάτων που θα κινηθούν με τα δικά τους μέσα δηλαδή για μια κατάσταση σαν startup κάτι που πρέπει να ελέγχεται ε, χωρίς μεγάλο διοικητικό άκτος αφού οι πόροι είναι χαμηλού ύψους πρέπει λοιπόν να, είμαστε, να δείξουμε περισσότερη επιμονή για αυτό το θέμα των αποτελεσμάτων, διότι αυτό που μετράει όταν επενδύουμε ευρωπαϊκά κονδύλια είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που θα ήθελα να μου πούνε επίση οι συναδέλφοι είναι θα μπορούσε ο καθένα με την εμπειρία του να βοηθήσουν ώστε να καθορίζουμε κάπω καλύτερα εφόσον επιτευχθεί το σωστό αποτέλεσμα να ε, απαλλασσόμαστε από την υποβολή επαχθών εκθέσεων, ε, οι οποίες είναι περιττές εφόσον έχει επιτευχθεί τόσο το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πολύ. Δεν βλέπω να επιθυμεί κάποιος όλος τον λόγο για να κάνει ερωτήσεις ή να σχολιάσει από τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζι. Δίνω τώρα το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Please. The floor is yours. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τα δικά σας σχόλια επί του θέματος. My name is Είμαι επικεφαλής της ομάδος για τη λειτουργική αποδοτικότητα στην ε, DigiRegio. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία της οργάνωσης αυτής της ε, ακρόασης για την απλοποίηση στα πλαίσια των θεμάτων περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ευρεία συζήτηση για το θέμα αυτό και όσο δυνατόν περισσότερους εμπλεκομένους για να μας δώσουν στοιχεία και συμβουλές για το θέμα αυτό. Αν μπορώ να ξεκινήσω με το να σταθώ σε ένα-δυο σημεία που ανέφεραν οι εμπειρογνώμονες μας στην αρχή. Ο Δόκτορης έκανε ορισμένε παρατηρήσεις σε σχέση με τον αριθμό των κατευθυντηρίων γραμμών και κανονισμών, τα έγγραφα, ο αριθμός των σελίδων σε κάθε έγγραφο. Αυτά είναι σωστά. Υπάρχει μεγάλο χαρτοβασίλειο. Γι' αυτό εγώ κυκλοφορώ με ένα iPad γιατί δεν τα βγάζω πέρα με όλα αυτά τα έγγραφα. Μόλον τούτο πρέπει να υπογραμμίσω ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτή την τεκμηρίωση γίνεται αιτήση των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε ό,τι αφορά για την κατεύθυνση καταρχήν. Εγώ είμαι υπεύθυνο για τον συντονισμό σε ό,τι αφορά τα έγγραφα αυτά στη γενική μου διεύθυνση. Αντίθετα από ό,τι πιστεύει ο πολλοί κόσμο, δεν το κάνουμε για πλάκα να έχουμε κατευθυντήρε γραμμέ και εγχειρίδια. Το κάνουμε μονάχα όταν μα το ζητούν. Στην Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, παραδείγματο χάρη, για την απλοποίηση ε, είχαμε, για το κόστος, είχαμε αυτήν την, ε, αυτό το εγχειρίδιο το οποίο είχε τόσο μεγάλο μήκος γιατί προσπαθούσαμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις των κρατών μελών και των διαφόρων αρχών για το απλοποιημένο υπολογισμό κόστους. Παρά τις προσπάθειές μας εξακολουθούν να μας πλημμυρίζουν ερωτήματα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και αυτό είναι μονάχα ένας μικρός τομέας του συνόλου της πολιτικής μας. Είμαστε καλοί υπάλληλοι της Κομισιόν, πρέπει να απαντήσουμε σε ό,τι ερώτημα και αυτό δημιουργεί ακόμα περισσότερα έγγραφα. Εδώ μπορείτε να δείτε μια <clears throat> συμβιωτική σχέση μεταξύ χαρτιού και ερωτήσεων. Όσο πιο πολλές ερωτήσεις, τόσο πιο πολύ χαρτί έχουμε. Και έχουμε φτάσει εδώ που είμαστε. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί για το θέμα αυτό μέσα στη χρονική περίοδο 2014-2020 δεν πρόκειται να ρίξουμε στην πυρά όλα αυτά τα έγγραφα που μας δίνουν οδηγίες για τα διαφορετικά ταμεία. Αυτό ίσως θα μπορεί να σκεφτεί το Κοινοβούλιο τι θα το κάνει, να το κάνει στο μέλλον μετά το 2020. Απλώς θέλω να εστιάσω σε αυτά που είπανε διάφορα μέλη της Επιτροπής σας σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε τώρα τι μπορούμε να επιτύχουμε σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Για μένα είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες απλοποίησης που περιλαμβάνονται ήδη στους κανονισμούς, στους κύριους κανονισμούς, στον κύριο κανονισμό, ο οποίος είναι ο κανονισμός CPR που έχει τις κοινέ πρόνοιες για τα περιφερειακά θέματα. Αν χρησιμοποιούμε όλοι το ίδιο ακρόνιμο θα είναι ήδη μια απλοποίηση να λέμε CPR λοιπόν, είπα ότι είναι πολλές οι δυνατότητες απλοποίησης, αλλά δεν υπάρχει καμία υποχρέωση απλοποίησης και αυτό είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για αυτούς τους κανονισμούς. Πολλοί εμπλεκόμενοι δεν θέλανε απλοποίηση, θέλανε ευκαμψία σε σχέση με τους κανονισμούς αυτούς. Η κυρία Καντέλα είπε κάτι πολύ σημαντικό, αναφερόμενη στο πρόγραμμα της απουλίας για την προσέγγιση <clears throat> με πολλά ταμεία, δηλαδή να είναι και το Περιφερειακό Ταμείο και το Κοινωνικό Ταμείο στον ίδιο κορβάνα. Πολλά κράτη-μέλη όμως δεν θέλησαν να ακολουθήσουν μια τέτοια απλοποιητική οδό. Αν μπορώ να σας παραθέσω τρία στοιχεία. Το απλοποιημένο κόστος είναι κάτι το οποίο το έχουμε ήδη αναφέρει. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό για να απλοποιήσουμε τη ζωή των προγραμμάτων και των δικαιούχων. Υπάρχει ένα α, κόστος το οποίο πρέπει να πληρώσει κανείς αν χρησιμοποιήσει την διαδικασία απλοποιημένου κόστους, θα πρέπει να έχουμε πρότυπο κόστος, να δούμε τι έχει γίνει ιστορικά για να μπορούμε να κάνουμε του υπολογισμούς για το μέλλον. Από τη στιγμή όμως που κάνουμε αυτή την προσπάθεια, από τη στιγμή που μιλάμε με τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τα συστήματα <clears throat> απλοποιημένου κόστους, ιδίως τα προγράμματα συνοχής, Όλοι αυτοί που έχω συναντήσει λένε τι ωραία που είναι, δεν θέλουμε να πάνε πίσω στο παρελθόν και να μην έχουν τη διαδικασία απλοποιημένου κόστους. Γι' αυτό η Γενική μας Διεύθυνση θέλει να προωθήσει το απλοποιημένο κόστος και η Επίτροπος Τάισεν παροτρύνει τις αρχές του Κοινωνικού Ταμείου στο να είναι τουλάχιστον τα μισά προγράμματα του κοινωνικού ταμείου μέσα από τη διαδικασία του απλοποιημένου κόστο και υπάρχει και μεγάλη λοκέρδο αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να πω, σε σχέση με το λογιστικό έλεγχο. Αν είναι απλοποιημένο το σύστημα κοστολόγηση, είναι πολύ πιο απλή και η διαδικασία λογιστικού ελέγχου. Μειώνεται τι ανάγκε για λογιστικό έλεγχο πολύ σημαντικά. Καταγράφω λοιπόν επίση αυτό που είπαν πολλοί ομιλητέ για τα θέματα του λογιστικού ελέγχου και του άχθου του λογιστικού ελέγχου πρέπει να πω ότι τα βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Καταλαβαίνω την ματέωση που νιώθετε, καταλαβαίνω τα σχόλιά σας για το άχθος που πρέπει να επομιστούμε, θα τα καταλάβαινα πολύ καλύτερα αν ο... ήταν καλύτερο το ποσοστό σφαλμάτων στην πολιτική συνοχή. Είναι πολύ δύσκολο να δικαιολογήσουμε το να γίνουν πιο απλές διαδικασίες και να μειωθούν οι λογιστικοί έλεγχοι όταν το ποσοστό σφαλμάτων στην, ε, στο Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχή είναι πολύ ψηλό. Αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε σε απλοποίηση. Και εδώ μπορεί να βοηθήσει η διαδικασία του απλοποιημένου κόστου. Τρίτο στοιχείο, γιατί το έθιξε κάποιο από του εμπειρογνώμονε, τα κοινά σχέδια δράση. Δεν υπάρχει κανένα τρόπο. Σε καμία περίπτωση ποτέ των ποτών που η Κομισιόν θα πάψει να χρησιμοποιεί τα κοινά σχέδια δράσης. Έχουμε εδώ εγχειρίδια που δίνουν κατευθύνσεις, λεπτομέρειες, επιλογές. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με τις εθνικές αρχές και τις διαχειριστικές υπηρεσίες για τη δημιουργία κοινών σχεδίων. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μάλλον απογοητευτεί από την έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των καθών μελών για τέτοια σχέδια. Αν είμαστε αισιόδοξοι θα λέγαμε ότι αυτό γίνεται γιατί έχουν εστιάσει στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων. Και τώρα που έχει περάσει αυτή, αυτή η πρώτη φάση θα υπάρξει περισσότερο ενδιαφέρον σε κοινέ δράσεις. Είμαστε έτοιμοι πάντως να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο γίνεται και περνάει από το χέρι μας. Η Επίτροπός μου, κυρία Κρέτσου, ανησυχεί πάρα πολύ για όλο το θέμα της απλοποίησης και ιδίω τον αντίκτυπο που θα έχει η απλοποίηση στους δικαιούχους. Γι' αυτό έχει πιέσει για τη δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επίπεδου για την απλοποίηση με την ε, με επικεφαλής τον πρώην Επίτροπο κ. Σιμ Κάλλας. Η ιδέα αυτής της ομάδας εργασίας είναι να εξετάσει τη, μια κέρια ομάδα από επιλογές ξεκινώντας με την έννοια του απλοποιημένου κόστους και της ηλεκτρονικής συνοχής και να δει πώς τα κράτη-μέλη, πώς τα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις βασικές ιδέες. Και όταν δεν τα χρησιμοποιούν τα προγράμματα, ούτε τα κρατημέλη, θέλουμε να τους ενθαρρύνουμε να το κάνουν, <clears throat> να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, να τις μεταλαμπαδεύσουμε όταν τα άλλα δεν ασχολούνται με αυτές τις πρακτικές και θέλω να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες μπροστά μας και είναι κέριο για την επιτυχία όλων των ευρωπαϊκών ταμείων διαφορετικού χαρακτήρα και επενδύσεων να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια και να τα κάνουμε πράγματι ελκυστικά για τους δικαιούχους να τα διεκδικήσουμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα εξασφαλίσουν με τη σειρά τους την επιτυχία της πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ πολύ ηχηρό το μήνυμα της Κομισιόν. Περνάμε στο τελευταίο μέρος της ακρόασης και της συζήτηση ε, και δίνουμε το λόγο στους ε, προσκεκλημένους, ε, τους εμπειρογνωμονές μας για να ακούσουμε κάποια τελικά οριστικά μηνύματα προς το ακροατήριο για τα διάφορα θέματα. Ξεκινάμε με τις κυρίες, κυρία Πετρέγγελ, ε, δύο-τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, όπως είπατε, ήταν ε, πολύ πλούσια η συζήτηση. Παρακολούθησα όλα τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας και χαίρομαι που ακούω ότι αρκετά από τα στοιχεία που ανέφερα εγώ νωρίτερα ε, έχουν απασχολήσει και σας και ειδικότερα κύριε Αλμπρεχτ είμαστε με το μέρο σας όταν ζητάτε για το μέλλον ένα ταμείο για να ευθυγραμμιστούν οι διευκαισίε και οι κανόνε. Αλλά ξέρετε, ο δρόμο προ κάτι τέτοιο ε, παραμένει δύσβατο. Ε, κάτι που μου προκαλεί ισοδοξία είναι ότι όλοι έχουμε ω κοινό στόχο τη μείωση του διοικητικού αχθούς ε, σε όλα τα επίπεδα ενδιαφερομένων αλλά ε, δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να βρούμε τον τρόπο. Πώς να το κάνουμε όλο αυτό, κύριε Ρόι, πρέπει να ε, έρθω σε επαφή με τους συναδέλφους μου στις διάφορες ενώσεις για να βρούμε γρήγορα διορθωτικά μέτρα, τρία γρήγορα διορθωτικά μέτρα όπως ζητήσατε. Αλλά ήδη αυτή η γράμμιση των ελέγχων είναι κάτι που όντως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί Επίσης και η καλύτερη σύνδεση με, τον, ε, με τη δέσμη μέτρων βελτίωσης της νομοθεσίας, το Better Regulation. Ε, στην Ευρώπη πρέπει να κάνουμε τις μειώσεις χωρίς να μπούμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες. Δηλαδή πρέπει ουσιαστικά να δούμε πώς αυτή η πρωτοβουλία Better Regulation, βελτίωση της νομοθεσίας, θα μπορούσε να βοηθήσει στην απλούστευση της πολιτικής ε, συνοχής ε, και ε, με τήρηση ταυτόχρονα των αρχών της. Αυτό που με ενθαρρύνει επίσης είναι αυτό που ακούσαμε από την Κομισιόν. Ειδικότερα για τα κοινά προγράμματα δράσης. Χαίρομαι που το άκουσα αυτό. Αλλά και για τις άλλες προτάσεις. Θα ρίξουμε μια ματιά και θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να σας κάνουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καντέλα. Λοιπόν, να επανέλθω στο ζήτημα του τι μπορούμε να κάνουμε όχι σε τρει μέρε, γιατί αν ήταν τόσο εύκολο, ε, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θα το είχαν ήδη κάνει. Τι μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες, γνωρίζοντας ότι έχουμε να κάνουμε με περισσότερα ταμεία, περισσότερα κονδύλια, ε, κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή αλλά υπάρχουν κάποια όρια μεταξύ όλων αυτών τα οποία θα έπρεπε να μπορούμε να υπερπηδήσουμε ώστε οι ενδιαφερόμενοι και οι αρμόδιοι υπεύθυνοι για την εφαρμογή ε, να μπορούν να εργάζονται μία φορά για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στον τομέα της κοινωνική καινοτομίας, ε, ο στόχος ανάπτυξης ε, επιτόπου ε, υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπου θα δοκιμάζουμε νέα μοντέλα υποδοχής με καταμερισμό χρόνου και υπηρεσιών. Πολύ ευρία έννοια φυσικά, εδώ αναφέρομαι σε αυτό που όλοι μας ονομάζουμε ε, ε, κοινωνική συστέγαση. Λοιπόν, για να τα κάνουμε όλα αυτά, με, να προσφέρουμε όλες αυτές τις διάφορες ε, δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να ζητούμε από τον υπεύθυνο εφαρμογής που θα είναι μία τοπική αρχή ή μια ένωση δήμων για παράδειγμα οι ιδιώτες ε, που είναι θεμελιώδη σημασία για να δώσουν περαιτέρω όθηση για την εφαρμογή μιας τέτοιας καινοτομία, μια πραγματικότητας για τη ζωή των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να τους ζητάμε να εργάζονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα με μερικούς διαφορετικούς στόχους. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ακόμη και το σύστημα των δικτών που μας προτείνουν οι κανονισμοί και που όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει για την αξιολόγηση των ε, επιχειρήσεων μας προγραμμάτων διαφέρουν μεταξύ τους. Σκεφτείτε το παράδειγμα της απολίας. Μία από τις λίγες περιφέρειες που αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την πολυτομιακή πολυταμιακή επιλογή. Εμείς βρεθήκαμε σε δύο διαφορετικά κομμάτια του ίδιου περιχειρησιακού προγράμματος να μιλάμε για το ίδιο πράγμα χρησιμοποιώντας διαφορετικούς δείκτες, ενώ μα εξυπηρετούσε η χρήση των ίδιων δικτών. Να σα δώσω ένα παράδειγμα, ένα πείραμα που κάναμε στο πλαίσιο του κύκλου 2007-2013. Σε αυτή τη δοκιμή το κάναμε άτυπα ουσιαστικά, off the record, χωρίς κανέναν ενδιαφερόμενο, ούτε χωρίς να λάβουμε υπόψη τους ελεγκτές, αξιολογήσαμε τις επιπτώσεις στην απασχόληση των ε, επενδύσεων του Περιφερειακού Ταμείου στις ε, κοινωνικές υποδομές σε εμάς. Εμείς αυτό το δίκτυο δεν μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε πουθενά. Δεν μπορούσαμε, δεν μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε πουθενά άλλου εκτός από την ίδια μας την περιοχή. Διότι το κοινωνικό ταμείο είναι ένας τομέας, ε, μου ζητούν βέβαια δείκτες ε, απασχόλησης, αλλά μόνο για τις δικές τους πολιτικές απασχόλησης. Αν δούμε τώρα το αποτέλεσμα και τα, τους πραγματικούς ανθρώπους που βρήκαν δουλειά, ε, χρειαζόμαστε μια προσέγγιση πολλών διαστάσεων όπως αυτή που χρησιμοποιούμε κατά τον προγραμματισμό. Τα παραδείγματα αυτά τι μας λένε ότι ε, πιθανότατα έτσι όπως έχουν τα πράγματα ε, ναι, απαιτείται χρήση πολλαπλών ταμείων, χρηματοδότηση πολλαπλών ταμείων, προγραμματισμό, σχεδιασμό των παρεμβάσεών μα. Αναπτύσσοντα εμεί λοιπόν ε, ενιαίου δείκτε αντί για έναν για τη μία γενική διεύθυνση και μία για την άλλη, μία για το ένα ταμείο και μία, ε, ένα δείκτη για το ένα ταμείο και ένα δείκτη για το άλλο, βοηθάμε και του υπευθύνου εφαρμογή να παρακολουθούν καλύτερα τα αποτελέσματα. Δεν θέλω βέβαια να περάσω εγώ κανένα μήνυμα μειώστε τους ελέγχους είναι πολύ. Αφού δεν ξεπερνάμε ένα ποσοστό σφάλματος και όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξυπηρετούν κάποιο σκοπό οι έλεγχοι. Αλλά πιστεύω ότι για να επιτευχθεί η απλούστευση αυτή τη στιγμή πρέπει να ε, μεριμνήσουμε για τους τρόπους με τους οποίους διενεργούνται οι έλεγχοι επί τόπου. Πρέπει να οργανώσουμε ολόκληρη την αλυσίδα, τη θεσμική αλυσίδα από τη διοικητική αρχή ξεκινώντας. Δεν βγάζω το, το, την τοπική διάσταση, δε, τους τοπικούς παράγοντες εκτός. Αυτό φυσικά είναι ένα κομμάτι της απλούστευσης. Δεν είναι μόνο ζήτημα κανόνων. Το πώς φτάνουν οι κανόνες μέχρι το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ε, ο τρόπο με τον οποίο φτάνουν μπορεί να βοηθήσει με κάποια σωστή οργάνωση των δραστηριοτήτων να μειωθούν τα κόστη. Α δούμε τη δειγματοληψία. Εμεί κάνουμε μια δειγματοληψία, μια άλλη δειγματοληψία κάνει η κυβέρνησή μα και άλλη κάνει η Κομισιόν. Και όπω συμβαίνει πολύ συχνά, ξαφνικά γίνονται ένα σωρό έλεγχοι. Ας μπούμε σε ένα χώρο μαζί και α κάνουμε τη δειγματοληψία μια φορά και α κάνουμε τον έλεγχο μια φορά, αντί να μαζεύουμε πληροφορίε από διαφόρου. Ε, ή να βάζουμε διάφορους να ζητούν από τον δικαιούχο ένα σωρό δείγματα και ένα σωρό ελέγχου. Σας το ζητάμε μια φορά, ας κάνουμε έναν έλεγχο πρώτου επίπεδου και ας βασίσουμε σε αυτό τους υπόλοιπους ελέγχους. Εμείς έχουμε αντιθέτως τρεις ανθρώπους που πάνε στην ίδια την ε, έδρα ε, στην έδρα της ίδιας επιχείρησης τρεις φορές για να στήσουν ακριβώς τα ίδια έγγραφα και σπάνια πάει να πει κάποιος δείξτε μου τις αίθουσες που διευθετήσατε Δείξτε μου τι έχετε κάνει στην πρακτική. Γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολη η συμμετοχή των διαφόρων παραγόντων. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δόκτωρ Ρης. Τα συμπεράσματά σας αν θέλετε, τα τελικά σας μηνύματα. Ευχαριστώ. Έχω να απαντήσω αυτό το ερώτημα από την βουλευτή της ε, Αυστρίας ποια είναι τα ωφέλη από αυτή την εναρμόνιση μεταξύ του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Αγροτικό Ταμείο Βέβαια Ανάπτυξης έρχεται από το Αγροτικό Ταμείο ε, Εγγύσεων. Είναι ένας άλλος κόσμος οριοθετημένος όπου υπάρχει ένας ε, έλεγχος των τρεχόντων δαπανών. Και έτσι λειτουργεί. Α, επίσης Έχουμε το πρόγραμμα Leader, το οποίο νιώθει μεγάλη υπερηφάνεια γιατί λειτουργεί εκ των κάτω προς τα πάνω. Και ενώ το, το Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Ταμείο θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, βλέπουμε ότι το Leader επιτυγχάνει χωρίς να γίνεται κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια γιατί βλέπουμε ότι εκεί έχουμε μικρές υποδομές. 60.000 ευρώ για μία μικρή υποδομή είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από τα κονδύλια που έχουμε στο Περιφερειακό Ταμείο και στο το Κοινωνικό Ταμείο που μιλάμε για δεκάδες εκατομμυρίων. Εγώ έχω ήδη πει ότι δεν είναι απαραίτητο να λειτουργεί η Κομισιόν με αυτόν τον τρόπο. Για μένα δεν πρόκειται να καταρρεύσουν όλα αν σταματήσει να λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Αλλά έχουμε τα κάτι μέλη που έρχονται στην Κομισιόν και λέμε μα φτιάξτε μας αυτό, κάντε μας εκείνο, κάντε μας το άλλο. Γι' αυτό έχουμε τις 60 σελίδες που θα πρέπει οι ελεγκτές να ελέγξουν. Αυτό είναι έγγραφο το οποίο προέρχεται από τους, ε, για τους ελέγχους. Σε με κάθε παραπάνω τεκμηρίωση αυξάνεται το ποσοστό των σφαλμάτων. Στο τοπικό μας ε, ελεκτικό συνέδριο του Λάντ μας ε, ελέγχθη το εξής για το Αγροτικό Ταμείο και για το Ταμείο Ανάπτυξης και το Ταμείο Εγγύσεων. Ακόμα και με δειγματοληπτικές ε, έρευνες δεν έχουμε ποτέ τη δυνατότητα να πετύχουμε να ελέγξουμε όλα αυτά. Έχουμε ακριβώς μόνο και μόνο με τις στιγματοληπτικές ε, έρευνες, με όλους αυτούς τους κανόνες, οι οποίοι οι ίδιοι δεν εφαρμόζονται σωστά, παράγεται ένα υπόβαθρο σφάλματων. Όταν έχουμε 60 σελίδες Έχουμε από τις 60 σελίδες 53 σελίδες από τα κράτη-μέλη και οι υπόλοιπε μονάχα είναι, σε, είναι πρωτοβουλία της Κομισιόν. Και να έρθω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το θέμα πάλι των λογιστικών ελέγχων. Όσο δεν έχουμε μια ενιαία διαδικασία λογιστικού ελέγχου, όσο δεν έχουμε ένα ενιαίο διοικητικό και ελεγκτικό σύστημα, ξεχάστε την έννοια των ολοκληρωμένων ταμείων. Το είπε η συνάδελφος από την Ιταλία. Όλα τα ελέγχουμε δύο και τρεις φορές. Εμείς έχουμε, τη, μπορώ να σας πω μια ιστοριούλα, μια περίπτωση που τη γνώρισα εγώ. Ήταν μια εταιρεία την οποία την ελέγξαμε εμείς και μετά ξανά ελέγχθηκε από ένα άλλο φορέα. Και αν μεταξύ έχει υπάρξει κάποιο σφάλμα, δεν μπορούμε εμείς να καταλαβαίνουμε τι γίνεται με το να έχει τα ίδια έγγραφα τα οποία, δηλαδή με το να πρέπει συνέχεια να παρουσιάζει διαφορετικά έγγραφα, παρουσιάζονται σφάλματα στο τέλος. Και τώρα, ο καθήτης Ντουγκάρο, τα τελικά σας σχόλια. Αυτός είναι τελός. Τελός, τελείως. Ευχαριστώ. Μεταξύ του 2000 και του 2015, Κάναμε ε, Κάνουμε μια γιγάντια λοιπόν προσπάθεια για την μείωση της εγγραφειοκρατίας. Για, αυτό, για αυτόν τον στόχο υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια επιτεύγματα, όμως η απλούστευση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το 2002 υπήρξε μία έρευνα της Eurostat Και εκεί ήταν ε, παρατηρήσαμε ότι υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων. Έπρεπε να ζητήσουμε τα πάντα από τους αρμόδιους υπουργούς του κάθε κράτους ε, μέλους. Έχει γίνει λοιπόν πρόεδρος από τότε. Μετά όσον αφορά την ε, συλλογή αυτών των μετρήσεων και την ένταξή τους στο, στις τελικές, στους τελικούς υπολογισμούς και εκεί ε, χωρίς τις, τα σωστά στοιχεία. Δεν μπορούμε να λάβουμε σωστές αποφάσεις. Η απλούστευση συμπεριλαμβάνει λοιπόν και αυτή την πτυχή. Αλλά αφήστε με να επιστρέψω στο πρόβλημα της ε, αποτελεσματικότητας. Προτού αναλύσουμε την απλούστευση της διαδικασίας, πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της απλούστευσης ε, αυτής. Διότι Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ε, που έχουν προταθεί για να βρεθεί λύση και ίσως συνδυάζοντα όλες αυτές να βρούμε μια κοινή κατεύθυνση, ε, διότι κάθε λύση είναι βασισμένη και σε ξεχωριστές προτεραιότητες και υπάρχει εδώ κίνδυνος ε, για πολλά επιχειρησιακά προγράμματα να αυξηθεί, να διπλασιαστεί ο φόρτος εργασίας. Η περιφέρεια της Τιμισοάρα της οποίας την στρατηγική επεξεργάστηκα, έχει πάνω από 300 διαμερίσματα, απασχολεί πάνω από 3.000 ε, υπαλλήλους. Εμείς δεν μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτού τους δείκτες ποιότητα, διότι δεν μπορούσαμε να, να φτάσουμε σε αυτού του δείκτες αποτελεσματικότητα που ε, προβλέπει αυτή η έξυπνη εξειδίκευση. Υπήρχε λοιπόν εμπόδιο αυτή εξ αρχή. Δεν ήταν το πρόβλημα λοιπόν η έλλειψη αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να καταλήξουμε. Κινδυνεύουμε να περιπλέξουμε τη διαδικασία υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Τα δεδομένα πρέπει να αφορούν, να, να αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, ενεργειακή ε, απόδοση κτηρίων. Υπάρχει μια αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία μπορούμε να βασιστούμε. Δεν ε, έχει νόημα να προσθέσουμε παράρτημα σε αυτήν την οδηγία, διότι έτσι περιπλέκονται τα πράγματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αρχική οδηγία για να φτάσουμε λοιπόν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Παράγεται ελάχιστη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία, το, η μεικτή προστιθέμενη αξία είναι 1,7% ανά κιλό, το πολύ 3,5% ανά κιλό ενέργειας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα έλεγα ότι μόνο μέσω της εξειδίκευσης και της έρευνας και της καινοτομίας θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε στον στόχο μας και πρέπει μην ξεχνάτε ταυτόχρονα να συνεργαστούν πολλές περιφέρειες μαζί. Μπορεί να υπάρχουν 15 περιφέρειες που θέλουν να φτάσουν στον ίδιο στόχο και χρειάζεται συνεργασία. Στον τομέα της ενέργειας, για παράδειγμα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο ε, πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Υπάρχουν οι τεχνολογίες εχμής, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, έτσι ώστε να είναι αποδοτικές. Όμως εδώ έχουμε το αντίθετο. Υπάρχουν πολλές μελέτες, ε, γίνονται πολλά έργα, όμως δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος διεξαγωγής των μετρήσεων. Ο κύριος Ευανίστελ Ρόι έκανε μια ερώτηση στην οποία μπορώ να απαντήσω κάπως γενικά. Σίγουρα μια ενισχυμένη προστιθέμενη αξία, μια αυξημένη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο και όχι μέτρηση μέσω του ΑΕΠ θα ήταν ένας Καλό σε δείκτης, θα ήταν μια καλή βάση για να αρχίσουμε, διότι έτσι μπορούμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα που ε, παράγεται σε κάθε περιφέρεια και θα λάβουμε υπόψη ε, μέσω αυτής της μεθόδου και τους μισθούς και άλλους δείκτες. Όμως ε, μόνο με την προστιθέμενη αξία δεν μπορούμε να είμαστε αρκετά σαφείς. Ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε σύγχυση, διότι πρέπει να υπολογιστούν πολλοί παράγοντες. Σίγουρα βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό η... να μειωθεί η κατανάλωση σε υλικούς πόρους γιατί υπάρχουν μελέτες, ε, γερμανικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι σε συγκεκριμένα υλικά, ότι για συγκεκριμένα υλικά οι πρώτες ύλες τελειώνουν. Σε 30-40 χρόνια θα έχουν εξαντληθεί και πρέπει λοιπόν αυτά τα αγαθά να παράγονται με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν αυτό είναι μια πτυχή της ε, αποτελεσματικότητας και πρέπει να δούμε πώς θα δαπανίσουμε χρήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τρίτον, στην Ευρώπη έχουμε εξαιρετικό εργατικό δυναμικό, εξαιρετικά καταρτισμένο. Είναι ένας φυσικός πόρος που πρέπει να εκμεταλλευτούμε εάν θέλουμε να ε, οδηγηθούμε σε αποτελέσματα τα οποία θα ωφελήσουν τους πολίτες. Υπάρχουν Υπάρχει αυτό το εξαιρετικό λοιπόν καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο δεν ε, χρησιμοποιείται επαρκώς από όλες ε, τις χώρες και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστούμε για την επικοδομητική συζήτηση αυτή, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε τους προσκεκλημένους μας. Πολύ ενδιαφέροντα τόσο μας είπαν, θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις μας και κλείνω αυτή τη συζήτηση και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης είναι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης της Επιτροπής Ρέτζι από το 2013 οι Επιτροπές ΕΚΟΝ και ε, ξεκίνησαν μια έκθεση ε, πρωτοβουλίας για την ΕΤΕΠ την έκθεση της ΕΤΕΠ για το 2014 ο ρόλος της ΕΤΕΠ για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω αφού η νέα γενιά πολιτικής συνοχής προβλέπει μεγαλύτερη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή μας αποφάσισε να καταρτήσει μια γνωμοδότηση για την ετήσια αυτή η έκθεση της ε, ΕΤΕΠ. Ε, προτείνω προθεσμία για τροπολογίες για αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση που θα συζητήσουμε σήμερα να είναι 12 το μεσημέρι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Προθεσμία τροπολογιών. Η συγκητής είναι ο κύριος Γιάκοφτσιτς, ο οποίος δεν είναι παρόν, οπότε επιτρέψτε μου εκ μέρους του να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης. Εκ μέρους λοιπόν του κυρίου Γιάκοφτσης, αγαπητοί συναδέλφοι, έλαβα ε, ειδοποίηση από τον κύριο Γιάκοφτσιτ ότι είναι ασθενή και δεν μπορεί να παρευρίσκεται στην απογευματινή μας συνάντηση. Έτσι λοιπόν μου ζήτησε να παρουσιάσω εκ μέρους του ορισμένα σημεία για αυτή τη γνωμοδότηση για την ετήσια έκθεση 2014 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επισημάνει τη σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων η οποία συμπληρώνει τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Ενώ πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και συγχρηματοδότησης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να παράσχει πολύτιμη υποστήριξη έτσι λοιπόν καλωσορίζει την αύξηση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ για το 2014 συμπεριλαμβανομένων άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ σε το δανεισμό και άνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ σε δρομολόγηση επενδύσεων που είναι ουσιαστική σημασία για τη συμπλήρωση της πολιτικής συνοχής καθώς και για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επένδυσης να τα συνεχόμενα προβλήματα όπως τα οικονομικά εμπόδια μπορώ να διακόψω. Το έχουμε. Ε, διαβάζετε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Το έχετε. Δεν θα το διαβάσω όλο, λέει η Πρόεδρος. Μπορώ να σας πω αυτή τη δική μου άποψη. Ε, αυτές εδώ είναι γραπτές σημειώσεις. Λοιπόν, τι πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Γιάκοψης εστιάστηκε στη θετική πτυχή της έκθεσης. Ανέφερε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τον ολένα αυξανόμενο ρόλο ουσιαστικά της τράπεζας και το δεύτερο κομμάτι της γνωμοδότησης ε, ε, αναφέρει επιλογές της, για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της ΕΤΕΠ και της Επιτροπής Ρέτζι. Αυτά είναι τα δύο σημεία που ήθελα να αναφέρω εγώ και σταματώ να διαβάζω το μήνυμα του κ. Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαν Εκτό. Εκτός. Είμαι σκιώδης του σκιώδους, ε, αναφέρει ο κύριος Βαν Και εσείς, του λέει ο πρόεδρος, σκιώδης του σκιώδους του σκιώδους. Λοιπόν, ξεκινάμε του σκιώδες. Κύριε Βαν Λίστεροι. Ε, κύριο Σίκλο για το Έλκδερ είναι εδώ, θα σας μεταφέρω το μήνυμά του και μια γενική παρατήρηση. Πιστεύω ότι η δομή της γνωμοδότησης είναι εντάξει. Αυτό που υπογραμμίσατε επίσης είναι η συνέργεια με τα δικά μας ταμεία και που πρέπει να υπάρχει. Όπως μόλις συζητήσαμε, ώστε να φέρει αποτελέσματα η περιφερειακή πολιτική μεγαλύτερα, μεγαλύτερες δηλαδή επενδύσεις από αυτές που έχουμε ήδη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά. Ο κ. Στίκο μου ζήτησε να υπογραμμίσω την υποστήριξη και για μικρότερα έργα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και όχι μόνο για τα μεγάλα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, περιλαμβάνει υπό την ίδια ομπρέλα και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και το υπογραμμίζουμε αυτό λόγω της έλλειψης ρευστότητας που χαρακτηρίζει αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η οποία τις οδηγεί σε προβλήματα επιβίωσης. Ε, τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν εισαχθεί θα βοηθήσουν αυτά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το άλλο σημείο αφορά την υποστήριξη που μπορεί να παράσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνεργασία με τους οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλοί άριθμα μέσα σε διάφορες χώρες και περιφέρειες, στα Λέντερ της Γερμανίας, που μπορούν να λειτουργήσουν ως ε, όχημα εξέλιξης. Αυτό καθίσταται δυνατό ήδη από το 2014 για να αναπτυχθούν οι δυνατότητες καινοτομία και μάθησης ώστε να γίνουν τα πράγματα σωστά, να μην γίνουν λάθη. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω επίσης ε, την σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, αν συνεργαστεί με αυτούς τους οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης ε, και τα σχετικά αυτά τα ταμεία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω φυσικά ότι ο κ. Γιακοφτσίτς έχει ζητήσει μακροπεριφερειακή στρατηγική και ειδική χρηματοδότηση για αυτή τη στρατηγική. Ε, μπορούμε να συμπεριλάβουμε και ένα σωρό άλλα πράγματα βέβαια. Ε, τις αναδυόμενες τεχνολογίες, ε, ε, βασικές τεχνολογίες, κέρυες τεχνολογίες όπως αναφέρονται στο νορίζοντα 2020, ε, όταν αναφερόμαστε τώρα ε, σε υψηλά ανταγωνιστικές νέες εξελίξεις ε, στα φωτονική και ένα σωρό άλλα πράγματα και εδώ ζητά συνέχιση της υποστήριξης των παραδοσιακών οικονομικών τομέων όπως γεωργίας, ναυπηγείων και τουρισμού ναυπηγική συγγνώμη και τουρισμού Αφού αναφέρουμε λοιπόν ορισμένου τομεί, πρέπει να αναφέρουμε και του πιο σύγχρονου τομεί που δημιουργούν θέσει εργασία. Πιστεύω. Αλλά εντάξει, θα φτιάξουμε κάποιε τροπολογίε για να υποστηρίξουμε ε, την γνωμοδότηση του κ. Κόφτσετ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρέσο, εξ του Σκιώδου των Σοσιαλιστών. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο. Έχει περάσει η ώρα, οπότε Ελάχιστε παρατηρήσει θα κάνω και μετά βέβαια ο ισχυρό συζητή μα θα διαβιβάσει το κείμενο στον εισηγητή. Ένα σχόλιο για να υπογραμμίσω το σημαντικό ρόλο της τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να προσφερθεί στις τοπικές αρχές. Διότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι η δυσκολία σχεδιασμού και προγραμματισμού με αποτέλεσμα προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότησης ή χρηστής αξιοποίησής τους. Η δεύτερη μου παρατηρήση σχετίζεται με την ε, ανάγκη που επισημαίνει και ο συνάδελφος να υπάρχει πιο στενή σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και ειδικότερα της Επιτροπής μας όσον αφορά τις κατευθύνσεις που ακολουθεί η ΕΤΕΠ για παρεμβάσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές υποδομές και ειδικότερα όπως ε, Αναφέρθηκε ήδη, υπενθύμψε ήδη ο συνάδελφος για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε κάπως να εμπλουτίσουμε το σημείο 8, το οποίο ήδη λαμβάνει υπόψη ο εισηγητής. Ε, τώρα πιο συγκεκριμένα μας δημιουργεί και τις αμφιβολίες το θέμα των οικονομικών ε, προσκομμάτων. Τι ακριβώς είναι, ε, θα θέλαμε να το διευκρινίζει καλύτερα ο εισηγητής στο κείμενο αυτό το θέμα των οικονομικών προσκομμάτων για να καταλαβαίνομαστε καλύτερα. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λούερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, συγγνώμη που έμπαινα και έβγαινα γιατί είμαι συντονιστή συγχρόνω σε δύο επιτροπέ. Δεν μπορώ να τι καλύπτω συνέχεια. Αυτή τη στιγμή ο Τζιμ Νίκολσον, φανταστείτε, και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάκοψης για τη γνωμοδότησή του. Υπάρχουν πολλές πτυχές που το ECR μπορεί να υποστηρίξει, ιδίως για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, η οποία θα υποστηρίξει τις επενδύσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα με τη διατύπωση στην αρχή της παραγραφού 8 που τονίζει τα, την προσέγγιση που βασίζεται σε αποτελέσματα για την πολιτική συνοχής στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 και τη συμβολή που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να αποδείξουμε στους φορολογούμενους μας λόγω της σημαντικής υποστήριξη στην πολιτική συνοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα χρήματα αυτά δαπανώνται με τρόπο σόφρονα. Σύμφωνα επίση και με τον εισηγητή για αυτά που λέει στο σημείο 2 και αναφέρθηκε και από άλλους αυτό ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα μεταξύ του ΕΦΣΥ, του Ταμείου Γιούνκερ και άλλων ταμείων. Πολλοί λοιπόν σε αυτή την αίθουσα θεωρούν ότι είναι πολύ αφηρημένο προς το παρόν το Ταμείο Γιούνκερ, το ΕΦΣΥ. Είναι μακριά κάπως ακόμα από τους δικαιούχους του. Αν μπορέσουμε να πτύχουμε λοιπόν μια καλύτερη σύνδεση μεταξύ του ΕΦΣΥ και του ESI, τότε μπορούμε σιγά σιγά να ξεπεράσουμε το αφηρημένο επίπεδο και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα του πόρου αυτού. Τέλο λέει ο Τζιμ. Ξέρω ότι η Επιτροπή Γεωργία θέλει να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να υπάρξει εξυγχρονισμό τη διαδικασία παραγωγή στο γαλακτοκομικό τομέα. Η Γεωργία είναι ένας τομέα όπου μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπογραμμίζω και πάλι ότι αυτή η δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων θα πρέπει να είναι συμβατή και συμπληρωματική με τις άλλες χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Σκλέρκ. Είστε και εσείς και ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Γιάκοτσης δεν είναι παρόν και θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω ιδιαίτερα θα ήθελα από τα εξής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να προωθήσει πολιτικές ε, περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την πλευρά των Πρασίνων θέλω να τονίσω ότι είναι σημαντικό να υπάρξει διαφάνεια στα χρηματοδοτικά μας εργαλεία και αναθεώρηση της λειτουργίας της. Το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο ανέφερε πρόσφατα ότι θέλει να διερευνήσει ένα, μάλλον υπάρχει ένα ενδεχόμενο σκάνδαλο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για εξαπάτηση από τη Volkswagen και υπάρχει το θέμα του αν αυτό το λογισμικό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι πληροφορίες επίσης για τους δικαιούχους είναι πολύ σημαντικό να είναι διαθέσιμοι. Το είπε και το ελεκτικό συνέδριο. Η έλλειψη πληροφοριών για τους τελικούς δικαιούχους έχει αρνητικά αποτελέσματα γιατί μπορεί να δημιουργηθεί η χρηματοδότηση αυτή και η καλύτερη σύνδεση με τους δικαιούχους για να δημιουργηθούν πράσινες θέσει εργασίας. Δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο και θέλω τελικά να αναφέρω ότι πρέπει να πληροφορούμε πάντως τους δικαιούχους για τις ευκαιρίες που έχουν για χρηματοδότηση και το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως αν έχουμε καθορίσει τους ε, ρόλους που θα πρέπει να ασκούνται από όλους εμπλεκομένους. Ευχαριστούμε ένας ακόμα, η κυρία Νταμάτο. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο, δεν είναι εδώ οπότε ε, δεν θα πάρω χρόνο τώρα για να εξοικονομήσουμε λίγο χρόνο. Ευχαριστώ. Ο εισηγητή λοιπόν και οι σκιώδε εισηγητέ φαντάζομαι ότι θα επεξεργαστούν το κείμενο και θα σα υπενθυμίσω η προθεσμία τροπολογιών είναι η Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Και τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα, ετήσια έκθεση 2014 για την υποστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολέμηση της απάτης. Βάσει του άρθρου 224 της Συνδίκης, Κομισιόν διατυπώνει μια έκθεση σε σχέση με τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουν το σεβασμό των οικονομικών συμφερόντων. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίσουν την απάτη. Αναφέρονται διαφορέ πολιτικέ όπω συγκεκριμένα και η πολιτική συνοχή. Εμεί ε, εκδίδουμε μια έκθεση πρωτοβουλία για το 2014 για τα θέματα αυτά. Ο εισηγητή μα είναι ο κύριο Βον, ο οποίο δεν μπορούσε να είναι παρόν σήμερα. Η κυρία Μπρέσο θα εκπροσωπήσει τον κύριο Βόν για την παρουσίαση της έκθεσης και σας υπενθυμίζω και πάλι ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι Τετάρτη 21 Οκτωβρίου δίνον τον λόγο στην κυρία Μπρέσου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα με τον κύριο Βόν δεν υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα σε αυτό το φάκελο παρότι τα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα. Όσον αφορά την πολιτική συνοχή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή δεν είναι ο τομέα με τον υψηλότερο αριθμό παρατυπιών. Στην πολιτική συνοχή οι περισσότερε παρατυπίε αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αν συγκρίνουμε τη σημερινή κατάσταση με το 2013, παρατηρείται αύξηση του 2% ε, στι παρατυπίες αυτό αντιστοιχεί σε 1.649 περιπτώσεις παρατυπιών που έχουν καταγγελθεί ως απάτες. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει κοινό ορισμός δόλων και μη δόλων ε, περιπτώσεων στην Ένωση. Διαφέρει ο ορισμός της απάτης ανακρατός και αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικά μέσα εντοπισμού των παρατυπιών και χρειάζεται να γίνει πιο ομοιόμορφο αυτό το σύνολο κανόνων διαφορετικά. Είναι αδύνατο να συγκρίνουμε τις, κατα... τις, καταστάσεις, το κάθε... τις καταστάσεις μεταξύ των κρατών μελών. Εμείς αναγνωρίζουμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά αυτές τις παρατυπίες και αναφέρεται μια ενδιάμεση αξιολόγηση στην έκθεση το 2018 που θα γίνει από εμά όπου θα αξιολογηθεί αν τα μέτρα της πολιτικής ε, συνοχής ε, καταπολεμούν την απάτη και μειώνουν τους κινδύνους παρατυπιών. Οπότε αναμένουμε εγώ είμαι εισηγητής και στην Επιτροπή ΑΦΚΟ για την ίδια έκθεση, εισηγητρία συγγνώμη. Πιστεύω ότι επίση θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να απλοποιήσει τη διαδικασία δημιουργώντα κατηγορίες, χωρίζοντας σε κατηγορίες ε, τα πιο τακτικά σφάλματα, τα πιο συχνά σφάλματα, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση μεταξύ σφάλματος και απάτης. Και ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα αποτελεσματικότερης καταπολέμησης των πραγματικών περιπτώσεων απάτης, ε, αντί να καταπολεμάμε σφάλματα, τα οποία ούτως άλλως μπορούν να αποφευχθούν. Αν ε, έχει οριστεί το συχνότερο σφάλμα με καθαρότητα και σαφήνεια. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλους σκιώδεις που θα ήθελα να πάρω το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι πλέον παράδοση να αντικαθιστούμε αλλήλους. Και έτσι λοιπόν και εγώ αντικαθιστώ το σκιώδη Γητή του ΑΕΛΚ. Γι' αυτό λοιπόν εξ ονόματός του θα ήθελα να πω τα ακόλουθα. Ή το... Για την πρόταση του κυρίου Βον. Λοιπόν, καταρχάς το ΕΛΚ θα ήθελα να τον ευχαριστήσει για την καλή τη δουλειά. Το σχέδιο έκθεσης είναι μια πάρα πολύ καλή αφετηρία για να αρχίσει η ανταλλαγή απόψεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το να υπάρξει απλοποίηση για εμάς, για το ΕΛΚΑ και είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν ε, είναι απαραίτητα όλα τα σφάλματα και περιπτώσεις απάτης. Χρειάζεται μία διαφοροποίηση, να ξεχωρίσουμε τα σφάλματα που έχουν γίνει χωρίς την πρόθεση απάτης και να δούμε πώς αυτά μπορούν να αποφευχθούν. Ωστόσο, το ΕΛΚ πιστεύει ότι Χρειάζεται απλούσταση και στη διαδικασία και στον κανονισμό, διότι αυτό θα συνεισφέρει στη μείωση του αριθμού σφαλμάτων. Οι δημόσιες ε, συμβάσεις είναι επίσης πολύ σημαντικό τομέα για το ΕΛΚ και αν δούμε την περιφερειακή πολιτική θα παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα κονδύλια πανώνται μέσω της διαδικασίας για τις δημόσιες προμήθειες ε, για, για τις κρατικές συμβάσεις. Αυτό λοιπόν υπάρχει ανάγκη απλούστασης εκεί έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση αυτών των λαθών. Και θα ήθελα εδώ να συστήσω στα κρατημέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις απάτης και να αντιδράσουμε σε αυτές. Και χρειάζεται επίσης να συμπεριληφθούν και οι αρχές και περιφερειακές αυτοδιοίκησης των αγώνων στο καταπολέμηση της απάτης και των σφαλμάτων. Ας μην ξεχνάμε ότι η απάτη αυτή ε, αποκτά όλο ένα και περισσότερο διεθνή χαρακτήρα, διασυνοριακό χαρακτήρα, γι' αυτό λοιπόν και χρειάζεται ανάληψη δράση σε διεθνές επίπεδο. Ίσως ε, να, θα, μπορούσαμε να συνεργαστούμε με την Γενική Εισαγγελία για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι αυτά είναι εν ε, ε, όσο ήθελε να πει το ΕΛΚ και είμαστε στην διάθεσή σας. Κύριε... Ευχαριστούμε κύριε Ντόιτζο. Κύριος Τσέζαρ, παρακαλώ. Πάνη Przewodnicząca, Szanowna Πάνη Przewodnicząca, ja w imieniu grupy EKR dziękuję Ευχαριστώ πολύ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της ομάδας των συντηρητικών θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση αυτή και να καλωσορίσω και όλα τα σχόλια των σχεδόν Είναι νομίζω η πρώτη γνωμοδότηση για την συγκεκριμένη περίοδο μέχρι το 2020 και πιστεύω πως χρειάζεται να τονίσουμε το ότι χρειάζονται αυτές οι αρχές, χρειάζονται αυτές ε, οι προτάσεις για την συνοχή και ότι πρέπει να γίνει κάτι διότι και από την πλευρά των δαπανών και από την πλευρά των εσόδων δεν έχουν σημειωθεί τόσο πολλά σφάλματα. Όμως, αν δούμε τα οικονομικά αποτελέσματα, θα δούμε ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό σφαλμάτων ε, κατά 6%. Αν δούμε επίση τις άμεσε ενισχύσει, ιδιαίτερα στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου, θα δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα κατάχρησης και απάτης σε ορισμένες ε, περιοχές. Τα τελευταία χρόνια και στα ταμεία συνοχής το μεγαλύτερο ποσοστό σφάλματος που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια ήταν 40%. Πρέπει να ερευνήσουμε την αιτία αυτών των σφαλμάτων και σε πολλές περιπτώσεις θα δούμε ότι πρόκειται για κατάχρηση των ταμείων και ε, κακή οικονομική διαχείριση. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένε περιπτώσει όπου τα ποσοστά ήταν πολύ ψηλότερα και πρέπει να δούμε, να αναγνωρίσουμε ότι αυτό είναι κάτι το ανησυχητικό, το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε στα πλαίσια των περιπτώσεων απάτη και σφάλματων. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας ε, δώσει κάποια στοιχεία για το γιατί αυξήθηκε αυξήθηκαν τα ποσοστά περιπτώσεων απάτης. Οι ελεκτές όταν ερωτήθηκαν για, τις, ε, για τους ελέγχους τους ε, στα πλαίσια της δαπάνης κονδυλίων από τα ταμεία αυτά, από τα κράτη-μέλη, μας είπαν ότι υπήρχαν περιπτώσεις ε, παρατυπιών, εισφαλμάτων ή απάτης αλλά ενδεχομένω να είχαν γίνει λάθη και είχαν όντω γίνει κάποια λάθη και ενδεχομένω να έχουν γίνει λάθη και σε άλλου τομείς. Πολύ συχνά τα σφάλματα αυτά έχουν να κάνουν με παρερμηνία των διατάξεων. Γι' αυτό πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εστιάσει στην βελτίωση αυτών. Επίσης, οι περισσότερες περιπτώσεις απάτης είναι τα παραποιημένα πιστοποιητικά Κάτι το οποίο έχει οδηγήσει φυσικά στην οικονομική απάτη, στη διαφθορά, στον τομέα αυτών. Όταν θέλει κάποιος να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και δεν ε, μπορεί, πολλές φορές ε, πλαστογραφεί έντυπα, παραπεί έντυπα. Χρειάζεται λοιπόν να διεξάγουμε τους ακατάλληλους αυστηρούς ελέγχους τόσο για να προλαμβάνονται τα σφάλματα αλλά και για να αποτρέπεται η απάτη. Πολλές φορές ίσως να χρειαστεί να οδηγηθούμε και σε αναστολή των ενισχύσεων. Εάν θέλουμε να κινητοποιήσουμε λοιπόν τη, τις προσπάθειες για τη μετώπιση αυτής της απάτης πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Χρειάζεται λοιπόν ε, μια υποχρέωση υποβολής ε, θέσεων, μια υποχρεωτική, ε, υποχρεωτική έλεγχη και οι κατάλληλοι μηχανισμοί για να καταπολεμήσουμε τις περιπτώσεις απάτης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέρκ. Έχετε το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αντικαστώ τον σκηριώδη μας εισηγητή και θα πω σύντομα Ποια είναι η θέση του σκιώδης συζητητή μας για την έκθεση αυτή. Χαιρετίζει την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για το 2014 σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των οικονομικών ε, συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν μπορεί να χαιρετήσει την έλλειψη πρόοδου σε σχέση με τις απάτες. Ανησυχούμε για το γεγονός ότι δεν έχουμε πληροφορίες για τις περιπτώσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί, το πώς οι περιπτώσεις αυτές συνδέονται με τα ποσά τα οποία ανακτήθηκαν. Υπάρχει ένα κενό χρονικό που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό το συσχετισμό. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε ένα σύστημα ε, ιχνηλασίας που μας επιτρέπει να ξέρουμε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι το συνολικό ποσό μετά από μερικά χρόνια. Τα ποσά θα πρέπει να μπορούν να συγκριθούν και να μπουν στο πλαίσιό τους, αλλιώ είναι περιορισμένα τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτά. Υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία όμως, δηλαδή χαιρετίζουμε αυτά τα οποία αναφέρονται στο, στην παράφορ 4 για τη συγκρισιμότητα. Μπορούμε να υποστηρίξουμε και αυτά που λέγονται για την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και διερεύνηση των συγκρούσεων συμφέροντος. Χαιρόμαστε λοιπόν και για το γεγονός ότι υπογραμμίζεται η σημασία της δημιουργίας ικανότητας και είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την διαφάνεια και την εταιρική σχέση για να μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία καλύτερα. Δεν βλέπω κανέναν σκιώδη πλέον. Ναι, ποιος, η κυρία Δαμάτο, όχι. Μου είπε όχι, ένευσε, αρνητικά. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από την ΟΛΑΦ εδώ, ναι. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Miss Maria... Η κυρία Μαρία Τσιόνι Γκόβας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο εισηγητή και όλα τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής σας ε, που αφιέρωσαν τόσο χρόνο για να μας ε, στείλουν κάποια σχόλια με αυτή τη, για αυτή την έκθεση έλαβα υπόψη και άκουσα όλα σας τα σχόλια. Θα τα λάβουμε υπόψη κατά την εκπόνηση της ε, έκθεσης της επόμενης, ε, αλλά επιτρέψτε μου κάποια σχόλια. Αναφέρατε και συγκρίνατε σφάλματα και περιπτώσεις απάτης. Θα ήθελα να σας πω ότι η έκθεση αυτή καταρχάς καλύπτει τις παρατυπίες και δόλιες παρατυπίες. δηλαδή υποψίες απάτης και διαπιστωμένες περιπτώσεις απάτης. Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις έχουμε πολύ σαφείς ορισμούς στο ενωσιακό, στο ενωσιακό δίκαιο και πρέπει να πω ότι αυτή η έκθεση δεν αναφέρεται σε σφάλματα. Ε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ε, και πρέπει να κάνουμε και τη σύγκριση με την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ μιας υπόθεσης που έχει αναφερθεί και του ποσού που έχει ανακτηθεί. Να υπενθυμίσουμε ότι στην κοινή διαχείριση η ανάκτηση αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους μέλους μεταξύ δικαιούχων. Ε, αληθεύει ότι σε επίπεδο επιτροπής έχουμε όλες τις πληροφορίες και κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα ε, στο πλαίσιο αυτής της σχέσης μεταξύ Επιτροπής και κράτους μέλους φυσικά για τις ε, υποθέσεις που έχουν αναφερθεί έχουμε κάποιες πληροφορίες στη βάση δεδομένων αλλά δεν πιστεύω ότι οι δικές μας πληροφορίες αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Γιατί, διότι τα ταμεία, η λειτουργία των ταμείων ε, της πολιτικής συνοχής όπως γνωρίζετε παρέχει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα όταν εντοπίζουν παρατυπίες πρώτα απ' όλα να τις διορθώνουν. Αυτό γίνεται βάσει του κανονισμού. Τι σημαίνει διόρθωση μέσω πιστοποίησης της δαπάνης Φυσικά σε επίπεδο κράτους μέλους υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης της ανάκτησης μέχρι επίπεδο δικαιούχου. Αλλά αυτό γίνεται μετά από, την, ε, από τον διακανονισμό μεταξύ κράτους μέλους και δικαιούχου. Something that uh, I really noticed. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση ήταν το θέμα βέβαια της διαφάνειας που επισημαίνεται και το θέμα της συνεργασίας με τους εταίρους, θα ήθελα να σας πω ότι εμείς στην Κομισιόν συνεργαζόμαστε φυσικά στενά μεταξύ μας εσωτερικά με τους διάφορους συναδέλφους, κυρίως στη Γενική Διευθύνση Περιφερειακής Ανάπτυξης και στη Γενική Διευθύνση Απασχόλησης, αλλά και με τα κράτη-μέλη. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε μία συνάντηση με τις υπηρεσίες ε, συντονισμού κατά καταπολέμησης απάτης στα κράτη-μέλη και συζητήσαμε όλα τα ζητήματα. Για παράδειγμα, 1η Δεκεμβρίου έχουμε συνάντηση με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες που είναι αρμόδιοι για τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. και μετά από τη δημοσίευση της δεσμής μέτρων για τις διατάξεις υποβολής εκθέσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο, μαζί με τα κράτη-μέλη θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε περαιτέρω το σύστημα υποβολής εκθέσεων, να ξεκαθαριστούν ουσιαστικά τα πράγματα και να λαμβάνονται άμεσα πληροφορίες από την Κομισιόν. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτά που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη, επειδή οι αυτέ καλύπτουν ε, κατά κύριο λόγο πληροφορίε, ενημέρωση βασικά προεκτέα από τα κράτη-μέλη, ε, εντοπισμό δηλαδή παρατυπιών. Οι πληροφορίε για την ανάκτηση ποσών σχετίζεται με την έκθεση Όλαφ. Αυτό σημαίνει έρευνα τη Όλαφ. Όπου φυσικά υπάρχει ίδια διαδικασία ανάκτηση, αλλά πρέπει να σα πω ότι η Κομισιόν δεν έχει ιδιαίτερε προφορίε ε, επ' αυτού ώστε να παρακολουθεί αυτού του είδου περιπτώσει. Ε, αυτά έχω να πω. Δεν ξέρω, Αντρέα, αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Σα ευχαριστώ πολύ, Λεκή Πρόεδρο. 21 Οκτωβρίου το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Περνάμε στο επόμενο θέμα τώρα. Το σχέδιο γνωμοδότησης για τις ε, συστάσεις προς το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις επί της Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών ΤΙΖΑ. Η, συγγήτρια μας είναι η κυρία Μόνικα Βάνα. Θα την αντικαταστήσει κάποιος, ο κύριος Κλέρκ, μάλιστα. Η συμφωνία αυτή για τις υπηρεσίες είναι υποδιαπεραγμάτευση από 25 μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, μέσα στους οποίους βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες αυτές καλύπτουν 70% του Παγκοσμίου Εμπορίου Υπηρεσιών. Η ΤΙΖΑ βασίζεται στη Γενική Συμφωνία για Εμπόριο και Υπηρεσίες του ΠΟΕ και έχει στόχο να ανοίξει τις αγορές στον τομέα των υπηρεσιών και να βοηθήσει την ανάπτυξη υπηρεσιών όπως είναι στην τηλεπικοινωνία χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και θαλάσσιες συγκοινωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται επί τη βάση της εντολής που της δόθηκαν τα 28 κράτη-μέλη του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο μπορεί να δεχτεί ή να απορρίψει τη συμφωνία, δεν μπορεί να την τροποποιήσει η Επιτροπή ΙΝΤΑ εκπονεί μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για να, καθα... να καθορίσει την άποψή της σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις γιατί αυτή η νέα συμφωνία μπορεί να έχει επιπτώσεις σε διάφορα επίπεδα και εμείς ε, θα κάνουμε αυτή την έκθεση ως Ρέτζι, θα κάνουμε μια γνωμοδότηση μάλλον στην έκθεση της ΙΝΤΑ για τις επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν σε περιφερειακό επίπεδο. 21 Οκτωβρίου είναι προθεσμία για τροπολογίες και πάλι την Τετάρτη την επόμενη και δίνω το λόγο στον κύριο Σκλέρκ, εξ ονόματος της κυρίας Βάνας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα μιλώ εκ μέρους της κυρίας Βάνα. Ε, έχει ανελειμμένες υποχρεώσει στη χώρα της και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Αποφασίσαμε ε, δυστυχώς ε, να διατηρήσουμε την ε, ώρα παρουσίασης αυτής παρότι είχε ζητήσει να συζητηθεί νωρίτερα. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς εκ μέρου της κυρίας Βάνα να σας ευχαριστήσω όλους και να σας ενημερώσω για το τι συμβαίνει ΤΙΣΑ είναι μια πολυμερής διαπραγμάτευση για την απελευθέρωση του εμπόριου των υπηρεσιών που άρχισε το Μάρτιο του 2013 και τώρα περιλαμβάνει 24 χώρες. Ο στόχος είναι η περαιτέρω ανα, ε, ανάπτυξη καλύτερων ασχέσεων και περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου των υπηρεσιών. Αυτή την εβδομάδα διεξήχθη ο 14 ο γύρος των διαπραγματεύσεων στην Γενέβη και το σχέδιο έκθεσης της ε, ε, Επιτροπή ΣΥΝΤΑ από την κυρία Ρέντινγκ ήταν έτοιμο επίση αυτήν την εβδομάδα. Υπήρξαν ορισμένε αλλαγέ σχετικά με τι αρμοδιότητε των τοπικών και περιφερειακών αρχών, την εξαίρεση δημόσιων υπηρεσιών κοινή ωφέλεια και κάποιε άλλε τώρα, γιατί χρειάζεται γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη. Το θέμα μας αφορά διότι η ΤΙΣΑ έχει επιπτώσεις ε, στις ε, δημόσιες συμβάσεις και το αποτέλεσμα των, ε, της συμφωνίας ε, ΤΙΣΑ θα έχει και επιπτώσεις στην ε, κοινωνική και, και περιφερειακή συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει το περιθώριο ελιγμών των πολιτών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών αλλά και της πολιτικής συνοχής θα επηρεαστεί. Γι' αυτό πρέπει να γίνει να γίνουν κατάλληλες διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να μην συμπεριληφθούν οι τοπικές, ή να μην συμπεριληφθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην συμφωνία αυτή. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τους ε, στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και ταφικής ε, συνοχής όταν θα, θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει για την συμφωνία ΤΙΣΑ. Αυτό που δεν θέλουμε είναι τα πρότυπα και οι αρχές της πολιτικής συνοχής να αποδυναμωθούν από την ΤΙΣΑ ή από οποιαδήποτε άλλη μελλοντική εμπορική συμφωνία. Θέλουμε οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να διατηρήσουν την αρμοδιότητά τους για την εφαρμογή όπως προβλέπει το άρθρο 1.3 της Συνδέκης του Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, των ε, διαφόρων επιμέρους διατάξεων. Τέλος, θέλουμε μια πλήρη εξαίρεση των δημόσιων υπηρεσιών από την Συμφωνία ΤΙΣΑ, κάτι που έχει εξάλλου ήδη προτείνει και η κυρία Ρέντινγκ. Επίση, κατά την κατάρτιση τη γνωμοδότηση, θα, κάποιες, θα προ, υποβάλουμε κάποιε τροπολογίε. Δυστυχώ, δεν είχαμε αρκετό χρόνο να υποβάλουμε τι ε, δικέ μα ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θέλαμε αυτό να τονιστεί στα πλαίσια της δημοκρατικής διαδικασίας. Επίσης, θα θέλαμε να ευαισθήσουμε την προσοχή στο ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν είχε αρκετό χρόνο να αντιδράσει. Επίσης, η κυρία Βάνα κλείνοντας ε, θα ήθελε να πει ότι θα χαρεί για τη μελλοντική συνεργασία με τους σκιώδες εισηγητές και για το αποτέλεσμα, δηλαδή την ε, γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Να σας ενημερώσω ότι δύο από τους σκιώδες εισηγητές ήδη έχουν στείλει στην κυρία Βάνα μία γραπτή ε, σε σχόλια, ο κύριος Πίκουλα από τους Σοσιαλδημοκράτες και ο κύριος Λούερ από τους ε, Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τάκουλα, τον σκιώδη συγητή των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, μπορώ να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα. Hyvät kollegat. Αξιότιμοι πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μερικές σκέψεις. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βάνα για τη δουλειά και τις προσπαθίες της και ο Σκιώδης ε, για το άλλο θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιες ιδέες. Η αρμοδιότητα τη Επιτροπής μας επί του ζητήματο αυτού είναι αμφισβητήσιμη, οπότε πιστεύω θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, κατά το χειρισμό αυτού του ζητήματος. Όσον αφορά το κείμενο της γνωμοδότησης, πιστεύω ότι γνωρίζουμε ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για ποιοτικά κριτήρια αναφέρεται σε ε, ανύψωση του επίπεδου των κριτηρίων και όχι υποβαθμισή του. Η Κομισιόν ε, έχει επισημάνει σαφώς ότι η υγεία, το περιβάλλον και τα λοιπά κριτήρια δεν θα αποδυναμωθούν. Μόνο θα ενισχυθούν. Επίσης πρέπει να σημειωθεί, αυτό πρέπει να επισημανθεί γιατί πρόκειται για μια γνωμοδότηση για ΤΙΣΑ. Αυτό δεν πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη συγκεκριμένη συμφωνία την οποία εξετάζουμε. Πιστεύω πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εντολή να αγγίξει τις δημόσιες υπηρεσίες στα κράτη-μέλη οι κυβερνήσεις των κρατών μελών είναι αρμόδιες να αποφασίζουν τι θεωρούν ότι είναι κρατικές υπηρεσίες ή δημόσιες υπηρεσίες. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια ώστε να μεριμνούν ότι οι περιφερειακές αρχές δεν θα ή τον βλάβη από αυτή τη συμφωνία. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δεχτεί το Συμβουλίο και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτή την πτυχή καθώς θα προχωράμε την εξέταση αυτής της έκθεσης. Πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή τη γνωμοδότηση, να λάβουμε υπόψη το στόχο της έκθεσης αυτής. Ο οποίος είναι μια ισορροπημένη συμφωνία που θα επιφέρει οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στα κράτη-μέλη. Θα χρειαστεί να κατανοήσουμε το μήνυμα που θα θέλει να στείλει η, Επιτροπή, η δική μας την Επιτροπή ΙΝΤΑ μέσω της γνωμοδότησης αυτής. Αυτές είναι οι απόψεις που ήθελα να μεταφέρω εδώ. Άκουσα ότι οι συναδέλφοι έχουν στείλει γραπτό στις απόψεις τους, το ίδιο θα πράξω και εγώ. Ώστε η εισηγήτρια να μάθει τις απόψεις μου. Είμαι βέβαιος ότι και ο συνάδελφος Κάρλεκ θα κάνει το ίδιο ε, για τις απόψεις που παρουσιάστηκαν εδώ σε αυτή τη συνάντηση και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε στο καλύτερη δυνατή λύση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νταμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο που επέμενε τόσο πολύ στην ανάγκη να εξεταστεί αυτή η γνωμοδότηση στη δική μας Επιτροπή. Θέλω να εκφράσω μία ανησυχία που θεωρώ δίκαιη και που επαναλαμβάνεται πολλές φορές στις παραγράφους του σχεδίου της έκθεσης. Η ανησυχία αυτή αφορά τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η ΤΙΖΑ στις αρμοδιότητες των περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά το η μυστικότητα που τις περιβάλλει, τις επιπτώσεις ε, για τις διάφορες περιοχές ή τις ε, ε, αναζωογονεί τις ανησυχίες μας όπως και η TTIP. Από τις πρώτες ειδήσει που έχουμε, από τα πρώτα νέα που έχουμε λάβει και από τα κείμενα των διαπραγματεύσεων, οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από διαφυγή εγγράφων, από δηλώσεις του Assange, που ήδη από καιρό έχει ε, δημοσιοποιήσει τα κομμάτια του ΤΙΖΑ που αφορούν τα οικονομικά. Διαβάζοντας κανείς το έγγραφο, θα ισχύει πέντε χρόνια μετά από την ε, σύναψη της συμφωνίας ε, ή αργότερα. Γιατί υπάρχει τέτοια μυστικότητα με αναφορά απλά στο απόρριτο των εμπορικών ε, ε, δραστηριοτήτων. Ε, πρόκειται να υπάρξει απελευθέρωση διαφόρων υπηρεσιών, μεταφόρων με μια ξέφρενη απελευθέρωση και αποτέλεσμα προβλήματα σε διάφορους οργανισμούς, σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορες αρχές και ειδικά περιφερειακούς και περιφερειακές και τοπικές αρχές. Μιλάμε λοιπόν για ουσιώδεις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι πολίτες μας καθημερινά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ε, υποβάθμιση των ουσιοδών αυτών υπηρεσιών προς όφελος των κερδών των συνήθων πολυεθνικών που μαζί με τις μειοπικές πολιτικές λιτότητες που ακολουθούν πολλές χώρες ε, οδηγούν στο λένε αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των ε, πλουσίων και των φτωχών σε πολλές ευρωπαϊκές κοινότητες. Όλο αυτό έρχεται σε αντίθεση με το στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που θα έπρεπε να επιδιώκει η εδαφική πολιτική και που εμείς εμβαθύνουμε στην Επιτροπή μας καθημερινά. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και Κωστέλο και μετά ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Ξέρουμε ότι όταν μιλάμε για μια παγκόσμια συμφωνία για το εμπόριο των υπηρεσιών, θα πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη προσοχή σε θέματα όπως είναι η προστασία των δεδομένων, η διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και η προστασία των δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Σας λέω ότι πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτά τα σημεία τα οποία μπορεί να είναι αμφιλεγόμενα, και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ανησυχίε γύρω από αυτέ. Θεωρώ, παρόλα αυτά, ότι αυτή η γνωμοδότηση όχι μονάχα θα πρέπει να σταθεί σε θέματα τα οποία είναι αρνητικού χαρακτήρα, θα πρέπει να αναφέρει και τα θέματα τα οποία έχουν θετικό χαρακτήρα, γιατί αυτή η Διεθνή Συμφωνία θα δημιουργήσει ευκαιρίες. Μπορεί με τον τρόπο αυτό να προωθήσει μια ενίσχυση και αύξηση της αγοράς υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα και επομένως με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Επομένως πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ των θετικών και αρνητικών. Εγώ δεν είμαι πάντα σίγουρος ότι μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα μονάχα με αρνητικό τρόπο. Θα πρέπει να κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία, λέει ο μιλητής, ώστε να δούμε και τις ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να προκύψουν από αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέγει πρόεδρος. Κύριε Λούερ, είπα ότι εστήλατε και μία γραπτή ε, συνεισφορά, αλλά θα θέλαμε να σας ακούσουμε και διαζώσεις. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά εδώ και θα ήθελα να πω κάπως ε, κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά, να εκφράσω την ευχαριστή προς την κυρία Βάνα για την έκθεση. Και εγώ ήθελα να πω ότι θα προτείνει να κάνουμε γνωμοδότηση εδώ στην Επιτροπή Ρέτζη. Αρχικά είχα σκεφτεί για ποιο λόγο να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τώρα αφού έχω σκεφτεί αντιλαμβάνομαι το πόσο ενδιαφέρον και το πόσο παρανοήσει δημιουργούν οι συζητήσει για τι εμπορικέ συμφωνίε με αποτέλεσμα διαρκείου διαλόγου. και για... Ε, χρειάζεται και περισσότερη διαφάνεια βέβαια, είναι σημαντικά χαρακτηριστικά αυτά. Επίσης αντιλαμβάνουμε πόσο σημαντικό είναι να άρουμε τα εμπορικά προσκόμματα στον όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο μας για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίω υπηρεσιών. Αντιστοιχούν σε κάθε εκατομμύρια θέσει εργασία ε, στον τομέα των υπηρεσιών στην Ευρώπη. Το να ανοίξουμε την αγορά σημαίνει αναμφίβολα μεγαλύτερη ανάπτυξη και θέσει εργασία. Α κοιτάξουμε την ιστορία. Οι άνθρωποι στη Βόρειο Κορέα ή στη Λευκορωσία ε, ζουν καλύτερα από ότι οι άνθρωποι στον Καναδά ή στη ΣΥΠΑ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στι κατοχώρε. Όχι βέβαια. Και υπάρχει λόγο. Ο λόγο είναι σαφή. Η συμφωνία τη ε, θα μπορέσει να αποδειχθεί πολύ σημαντική θα δώσει όθηση 20 δισεκατομμυρίων λιρών Αγγλίας στο ετήσιο ΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μεγαλύτερο το ποσό από τη συμφωνία, αυτό παρέχει η συμφωνία με τον Καναδά. Θα ωφελήσει τις ε, επιχειρήσεις στο χρηματοπιστωτικό, στο ψηφιακό τομέα, στις τηλεπικοινωνίες, στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Είναι πράγματι ένας από τους ε, βασικούς λόγους που εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούμε να υποστηρίξουμε τη συνέχιση τη ιδιότητας μέλους μας. Η αύξηση λοιπόν της διαφάνεια θα μπορέσει να υποστηρίξει το ευρύτερο θεματολόγιο τη ενίας αγορά στην Ευρώπη. Ακόμη και η κυρία Ρέντινγκ, ε, η συγκίτρια της ΙΝΤΑ, ανέφερε στο έγγραφό τη ότι αφού ο κόσμος δεν γνωρίζει πια σύνορα και οι κανόνες δεν πρέπει να γνωρίζουν σύνορα και η απελευθέρωση αυτή των υπηρεσιών ε, πρέπει να γίνει γιατί είναι μεγάλα τα προσκόμματα μεταξύ των χωρών. Ε, ωστόσο πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα πρότυπα θα περιμένουν υψηλά και ότι οι αρχές θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται τις δημόσιες υπηρεσίες όπως θεωρούν κατάλληλο. Έτσι λοιπόν υποστηρίζουμε τους στόχους, την ενίσχυση των προτύπων και τη δημιουργία ενός πιο ανοιχτού και ε, χώρου ανταγωνισμού όταν οι δικές μας εταιρείε ε, δραστηριοποιούνται σε άλλες Πιστεύω ότι θα μπορέσουν μπορέσουμε, ε, πιστεύω ότι θα μπορέσω να υποβάλω τροπολογίες τέτοιες που θα λάβουν την υποστήριξη των περισσότερων συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την συζήτηση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 21η Οκτωβρίου, Τετάρτη. Και εδώ Ολοκληρώσαμε τα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης μας για σήμερα. Πρέπει τώρα να εγκριθούν οι αποφάσεις των συντονιστών. Να σας πω ότι συνεδρίασαν νωρίτερα σήμερα οι συντονιστές και οι αποφάσεις τους έχουν σταλεί σε όλους σας. Υπάρχουν σχόλια, συμφωνείτε. Κύριε Βανίστε, Λερόι. Ναι, θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά στο κείμενο, ε, γιατί έχω δύο μικρές παρατηρήσεις. Καταρχάς, ας μην παρεξηγηθώ, οι προφορικές ερωτήσεις δεν ε, είναι ε, όλες ερωτήσεις ε, όπου είμαστε σύμφωνοι. Συμφωνούμε μόνο σε τρεις από αυτές. Έχουμε συμφωνήσει να εθετήσουμε μία προσέγγιση βήμα-βήμα. Σχετικά με την απλούστευση, εμείς είμαστε τρίτη στη σειρά. Έπειτα, σχετικά με την απόφαση για τον ορισμό εισηγητή για την Ελλάδα, για τον μόνιμο εισηγητή. Να σας πω ότι πήραμε την απόφαση να τον ονομάσουμε μόνιμο εισηγητή για να μην ε, δημιουργηθεί σύγχυση με τους ε, συνηθείς εισηγητές εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι δεν πρόκειται για την ε, συνηθισμένη ιδιότητα του εισηγητή. Πρόκειται για μόνιμο εισηγητή, standing reporter και αυτή την ορολογία θα χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα. Να σας ενημερώσω ε, για το ότι οι προφορικές ερωτήσεις έχουν ήδη, όπως τα λέγω, ήδη βάλει την υπογραφή μου στην επιστολή σχετικά με τις προφορικές ερωτήσεις. Φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά τους για να δείξουμε την σημασία που έχουν και την προτεραιότητα που έχει κάθε προφορική ερώτηση για εμάς. Σας παρακαλώ. Επίσης, να σημειώσουμε τον μόνιμο εισηγητή, αυτήν την ιδιότητα του μόνιμου εισηγητή. Ωραία, λοιπόν, ολοκληρώσαμε και εδώ τι αποφάσει των συντονιστών. Υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Τίποτα. Περίμενα να έχουμε έναν μακρύ κατάλογο για τα διάφορα, αλλά όχι. Επόμενη συνεδρίαση 12 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις μισή το απόγευμα. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τους διερμηνείς για τη βοήθειά τους σήμερα αυτή την μεγάλη μέρα που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ Λία τη συνεδρίαση.